Colleagues, good morning. Καλημέρα, συνάδελφοι. Ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση, ανακοινώσεις του Προέδρου, καθορισμό εισηγητών, συντακτών, κειμένων. Τι αποφάσισαν οι συντονιστές στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις τους τώρα εισηγητέ και συντάκτες κειμένων. Δύο εκθέσεις έχουν κατανεμηθεί. Η Σύμβαση των Αθηνών για, το, για τους επιβάτες ε, ζητήθηκε από το Συμβουλίο σαν αφορά την προσχώρηση του Ευρωπαϊκής Ενώσεως το πρώτο 2002 και απόφαση των συντονιστών είναι να ανατεθεί στον Πρόεδρο ή όποιος θα καθοριστεί να το κάνει. Δεύτερον, έχουμε τη γνωμοδότηση για οδηγίε όσον αφορά τη χρήση των PNR, των αρχείων επιβατών, στοιχεία για πρόληψη, έρευνα, εντοπισμό και δίωξη τρομοκρατικών ε, δικημάτων, σοβαρών εγκλημάτων. Αυτή είναι η γνωμοδότηση. Πηγαίνει στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, νομίζω. τους πρασίνους, διότι οι πράσινοι είναι οι επόμενοι που έχουν σειρά, οπότε οι πράσινοι μπορούν να μας γνωστοποιήσουν ποιος θα τον Μπορούμε να μαντέψουμε, αν μπορείτε επίσημα να μας πείτε, θα σας είμαι θα ευγνώμονες. Και για τα έγγραφα προς ενημέρωση, έχουμε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενδιάμεση αξιολόγηση της ε, σύμπραξης ΕΖΑΡ ε, και συμφώνησαν οι συντονιστές με την πρόταση να καλέσουμε τον Διευθυντή του ΣΕΖΑΡ σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις της ε, Επιτροπής μας. Τέλος, όσον αφορά τις συμφωνίες για αερομεταφορές και εμπιστευτικά έγγραφα, οι συντονιστές συμφώνησαν λογικό κώδικα πρακτικής που θα πρέπει να εφαρμοστεί σύμφωνα με την προσέγγιση που ακολουθήθηκε στην επιστολή που έστειλε υποφαινόμενος και επίτροπος Κάλλας και θα ήθελα απλώ να σα ενημερώσω επ' αυτού, γι' αυτό σα αναφέρω. Και τέλο, οι συντονιστέ μου ζήτησαν να στείλω σχέδιο επιστολή στον κύριο Μπαρόσο σχετικά με δημοσιονομικούς πόρους για πολιτική σχετικά με τον τουρισμό. Αυτή η επιστολή απεστάλλει. Οπότε ε, στρέφομαι προς τις χθεσινές αποφάσεις των συντονιστών. Όσον αφορά την ομάδα, υψηλή ομάδα συντονισμού ε, για τη ΣΤΟΑ, και το βραβείο για τη βιώσιμη ενέργεια πρότειναν οι συντονιστές η κυρία Τσίκαου επειδή είναι παλιά πρόσωπο της ΣΤΟΑ να εκπροσωπεί τη ΣΤΟΑ στην ομάδα υψηλού επίπεδου συντονισμού ε, για την επιτροπολογία και εδώ περιπλέκονται κάπως τα πράγματα συνάδελφοι οπότε προσέξτε με και δείξτε υπομονή ο Πρόεδρο ενημέρωσε του συντονιστέ για μια συνεδρίαση των εμπειρογνωμόνων δυνάμει του άρθρου 15 τη Συμφωνία Πλαισίου, ε, συναντήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συναντάται με εθνικού εμπειρογνώμονε για την ετοιμασία και εφαρμογή ε, νομοθεσία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να καλεί εμπειρογνώμονε του Κοινοβουλίου επίση, αν το Κοινοβούλιο ε, θέλει κάτι τέτοιο. Εγώ αντάλλαξα σχετικά επιστολές με τον Αντιπρόεδρο Κάλλας σχετικά με την οδηγία ITS όπου η Επιτροπή Μεταφορών ίσως ζητήσει να είναι παρούσα και η πρώτη συνεδρίαση προβλέπεται το μήνα Μάιο. Δεν υπάρχουν προσανατολισμοί ποιοι θα είναι οι εμπειρογνώμονε του Κοινοβουλίου. Αυτή τη στιγμή συμφώνησαν τα εξή οι συντονιστέ να σα προτείνουν. Το Κοινοβούλιο μπορεί να εκπροσωπείται όταν είναι αναγκαίο από τον Πρόεδρο, ο οποίο θα παρίσταται, παρακολουθεί τι συναντήσει και από τον εισηγητή. Μπορεί ο πρόεδρο να αναθέτει την εποπτεία του σαν αντιπρόεδρο ή το μόνιμο ε, εισηγητή για την επιτροπολογία. Ένα μέλο τη γραμματείας θα πρέπει να πάρει στι συνεδριάσει για την προετοιμασία, το κατεξιδότηση πράξεων και σε συνεδριάσει εμπειρογνωμόνων χρειάζεται και να ενημερώνει ε, σχετικά τα μέλη και να απευθύνει προσκλήσει για τι συνεδριάσει. Αυτή είναι η πρόταση λοιπόν η σύσταση των συντονιστών. Όσον αφορά το διαθρωμένο διάλογο, το διάλογο, ο Πρόεδρος να υπενθυμίσει ότι η προθεσμία για ε, συμμετοχή των πολιτικών ομάδων για το πρόγραμμα εργασίας ε, για το 2012 είναι 30 Μαρτίου και θα πρέπει να συμφωνήσουμε πάνω σε 4 με 6 προτεραιότητες από το πρόγραμμα εργασίας. Μία προτεραιότητα θα είναι υπερπροτεραιότητα, υπαριθμόν ένα προτεραιότητα. Και οι συντονιστές ε, θα ε, συζητήσουν στις 11 Απριλίου αυτές τις προτεραιότητες. Στα διάφορα ο Πρόεδρο ενημέρωσε τους συντονιστέ περί ενδεχόμενη συνεδριάσεως που θα μπορούσε να συγκληθεί συνάντηση μεταξύ αυτών και του κυρίου Κάλλα για τη Λευκή Βίβλο πριν δημοσιευτεί αυτή η βίβλο επισήμω, για την επίσκεψη στην προσωπή στο Μαρόκο ο μέγιστος αριθμός θέσεων είναι 8 μέλη για την επίσκεψη στο Μαρόκο διότι είναι επίσκεψη εκτό Ευρωπαϊκή Ενώσης σύμφωνα με τον ΤΕΟΝΤ ο καθορισμός θέσεων είναι 4 για το ΕΛΚ, δύο για το SND, μία ALDE και μία ECR. Τώρα και κλεισμένο το συνάντηση με τον νέο διευθυντή, για τον κύριο Baldwin, για τι αερομεταφορές. Είναι σήμερα στις 5 και 30. Να υπενθυμίσω στα μέλη ότι είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα συνεδρίαση και οι συγητές και σκιώδεις προσεκλήθησαν μαζί με του ε, συντονιστέ η παρουσία των πολιτικών ομάδων, των προσωπικού των πολιτικών ομάδων που περιοριστεί σε δύο μέλη, οι σύμβουλοι κατά ομάδα και βοηθή μελών ένα άτομο κατά μέλος αν θέλουν να παρίστανται και τέλος να υπενθυμίσω ότι η συνεδρίαση της Επιτροπής τον Απρίλιο θα λάβει η χώρα στις 13 Απριλίου το πρωί, μάλλον ακυρώνεται. Η πρωινή συνεδρίαση στις 13 Απριλίου συστήνεται, προτείνεται να ακυρωθεί. Αυτά έχω να πω όσον αφορά τους συντονιστές. Έχετε σχόλια, ερωτήσεις σχετικά με αυτά που σας είπα. Αν δεν έχετε, μπορούμε να συμφωνήσουμε λοιπόν όσον αφορά τις πληροφορίες και τις ανακοινώσεις που σας έκανα. Σας ευχαριστώ λοιπόν γι' αυτό. Μπορούμε να προχωρήσουμε και να πάμε στις ψηφοφορίες. Συνάδελφοι, πολλή κουβεντούλα γίνεται, μπορούμε να ησυχάσουμε λίγο να μιλάτε πιο χαμηλόφωνα αν έχει την καλοσύνη. Πρώτη ψηφοφορία, η έκθεση της κυρίας Τσικάου όσον αφορά την εφαρμογή του δορυφορικού συστήματος πλοήγησης του παγκοσμίου αυτού συστήματος. Πριν ξεκινήσουμε, ας κάνουμε μια δοκιμή, μια δοκιμή ψηφοφορίας, πρακτική αν θέλετε. Ξεκινάμε αυτή τη δοκιμή μας. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Όλα καλά, κυρία Κάστονιτς. Όλοι ψήφισαν. Αυτοί που έπρεπε να ψηφίσουν ψήφισαν και όχι παραπάνω. Έχετε όλοι τις κάρτες σας. Ωραία. Ξεκινάμε με την έκθεση κυρία Τσικάου Παράγραφος 2 λοιπόν, τροπολογία 13 της κυρίας Λίχτενμπέργκερ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ. 14 του κύριου Κούν. Κατά αποχές εγκρίνεται 15 με προφορική τροπολογία αντικαθαστεί η ΕΑΣΑ με αρχές. Έχουμε αντίρρηση αφορά την προφορική τροπολογία. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, ψηφίζουμε αυτή την προσφορική τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 16 κουν υπέρ. Κατά απόχέ, εγκρίνεται. 17 Μαρινέσκου υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 5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 αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 προφορική τροπολογία που αφορά την παράγραφο 11, συμβιβαστική 2. Δεν είμαι σίγουρος που μπορεί να έχουμε συμβιβασμό προφορική τροπολογία, αλλά τι να κάνουμε, αυτό έχουμε. Υποθέτω ότι δεν υπάρχουν αντιρρήσεις αφορά την προφορική τροπολογία. Συμβιβαστική 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 43 και κόζα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράθεση 2α1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 2 ουτζίας με προφορική τροπολογία Είσαστε όλοι ικανοποιημένοι με τροπολογία την προφορική υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. τρία; υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. τέσσερα; υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. έξι με προφορική τροπολογία. Είσαστε ικανοποιημένοι με αυτήν. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται.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 κατά εποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καλώς τελική ψηφοφορία που ξεκινάει. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Okay. So Ευχαριστώ. Σημειώνω ότι είσαστε υπέρ. Λοιπόν, 38 ψηφίσαντε συν έναν, 39 με τον κύριο Πασκό. 30 υπέρ, 1 κατά και 4 αποχέ. Εγκρίνεται λοιπόν συγχαρητήρια στην εισηγήτρια την κυρία Τικάου. Can I go on now to my own... Να περάσω στη δική μου έκθεση τώρα αν μου επιτρέπετε. Λοιπόν, τροπολογία 2, runner, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3, Μάιστινερ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4, με μια προφορική τροπολογία αν συμφωνείτε. Ωραία, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πέντε, Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έξι, Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Επτά, Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9. Τεφέρακ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8. Λίχτεμπεργκε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12 καταπίπτει. Παράγραφος 14 μια προφορική τροπολογία των σοσιαλιστών. Αν συμφωνείτε, υπέρ, κατά, απαχές, εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, απαχές, εγκρίνεται. 15 με την προφορική τροπολογία. Αν συμφωνείτε, ωραία υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται και ένα runner υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά άρχεται. Just keep your thumb up, Mr. Tapaski, Those, everybody voted. The vote is closed. Πέρας ψηφοφορία. 39 ψηφίσαντε με τον κύριο Πάσκο και 39 υπέρ. Καμία αποχή. Εγκρίνεται. Δεν λέω συγχαρητήρια τότε στον εισηγητή ή να πω. Οκ. Okay. Καλώς. Επόμενη. Έκθεση σε Νάλοβα για την οδηγία του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου που τροπολογεί το 2025 για τους ελκυστήρες που υπάρχουν στην αγορά μας στα πλαίσια του ευελικτού συστήματος. Πέντε τροπολογίες. Τροπολογία 1 Λίχτενμπεργκ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τρία. υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 3. Άρχιδη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 18 υπέρ, 19 κατά. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται. As everybody voted. Ψήσαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 39 ψηφίσαντε, 31 υπέρ, 4 κατά, 4 αποχές. Συγχαρητήρια στην εισηγητήρια κυρία Συνάλογα. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης που είναι η Ευρωβινιέτα, επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά. Ο κύριος Αλκαντράου έχει το λόγο. Dank u wel, voorzitter. Ik zou om te beginnen de, de schaduwrapporteurs en de verschillende fracties willen danken voor de... Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους σκιώδεις συγητές για την ε, αγαστή συνεργασία που είχαμε τις τελευταίες εβδομάδες. Ε, επιτρέπουμε με την οδηγία αυτή στα κράτη-μέλη, αν το επιθυμούν, να χρεώσουν τους οδικούς χρήσης και με εξωτερικό κόστος και εξασφαλίζουμε μεγαλύτερη ελαστικότητα για τα κράτη-μέλη. Έτσι θα προκύψουν κάποια κονδύλια που θα μπορέσουν τα κράτη-μέλη να τα επενεπενδύσουν στους τομείς των μεταφορών ώστε να εξασφαλίσουν κάποια μεγαλύτερη βιωσιμότητά τους. Επίσης, επιχειρούμε καλύτερο συντονισμό και σύγκληση μεταξύ μας για να συνεχίσουμε στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Ας μην ξεχνούμε ότι στη δεύτερη ανάγνωση δεν μπορούμε να απορρίψουμε τη θέση του Συμβουλίου, απλώς να τη βελτιώσουμε, να την διευκρινίσουμε, να τη συγκεκριμενοποιήσουμε και απαιτείται γι' αυτό ειδική πλειοψηφία. Ως εισηγητής και από την αρχή της προσπάθειάς μου, προσπάθησα να καταρτήσω μία σειρά τροπολογιών που θα αποτελέσουν την καλύτερη δυνατή φάση, βάση για τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και θα συσπηρώσουν όσο το δυνατό περισσότερους συναδέλφους. Και μάλιστα στις συμβαστικές αυτοστροπολογίες προσπάθησα να λάβω υπόψη τις ανησυχίες των συναδέλφων και όχι να περιλάβω τις δικές μου απόψεις που μερικές φορές ήταν πιο φιλόδοξες. Μιλάω για τη διαλειτουργικότητα, την ανάγκη καλύτερου, καλύτερης αναρμόνισης των μεθόδων υπολογισμού και επίση επικεντρώθηκε στην ανάλυση πέντε σημείων. Καταρχήν, η επιλογή του εξωτερικού κόστου ε, που θα καταλογιστεί στο μέλλον. Όλα αυτά μπορούν να εξεταστούν στο πλαίσιο της δυνατότητας ε, καλύτερης εφαρμογής ε, των υποδομών για την ίσπραξη των τελών. Επίσης ασχολήθηκα ιδιαίτερα με το θέμα της επιλογής του εξωτερικού κόστους που λαμβάνεται υπόψη. Για μένα είναι θεμελιώδες αυτό το ζήτημα. Και επίσης ε, τα έσομαι και εγώ υπέρ μια διαφοροποίησης, όπως και το Συμβούλιο αυτού του εξωτερικού κόστους. Δίνω έμφαση και στο θέμα της ουδετερότητα αυτής της προσέγγιση, τη δημοσιονομική ουδετερότητα και προσπάθησα να το διευκρινίσω. Η διαφοροποίηση θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό μεγαλύτερη γίνεται, να υπερβαίνει ακόμη και το 200% των μέχρι τώρα ποσών που προτάθηκαν. Επίσης, λαμβάνουμε υπόψη τι θα πρέπει να γίνει στις ε, περιόδους εχμής. Το Συμβούλιο πρότεινε 5 ώρες, εμείς προτείναμε 8, αλλά είναι υποδιαπραγμάτευση και αυτό το θέμα. Με την προσέγγιση αυτή νομίζω ότι προσαρμοζόμαστε καλύτερα στην πραγματικότητα σε ορισμένες περιοχές της Ένωσης, που μερικές φορές οι περίοδοι εχμής αγγίζουν και το οκτάωρο. Και το θέμα της προσημής, του προκαθορισμού των κονδύλιων. Να προβλέψουμε δηλαδή που θα χρησιμοποιηθούν. Το 2006 ήδη είχαμε ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Η θέση του Συμβουλίου εδώ είναι σαφής. Μας λέει δηλαδή το Συμβούλιο ότι θα λάβει υπόψη κάποιες συστάσεις για την επανεπένδυση των κονδυλίων, των εσόδων που συγκεντρώθηκαν στο, στις μεταφορές, αλλά εμείς θέλουμε να μην είναι προαιρετική αυτή η επανεπένδυση, αλλά υποχρεωτική, δηλαδή οπωσδήποτε αυτά τα έσοδα να επαναεπενδύονται στις μεταφορές. Και αυτή θα είναι η θέση μας στο Συμβούλιο, ενώ το Συμβούλιο προτιμά μια φαιά ζώνη που θα ευνοεί τους πάντες. Μία άλλη απέτησή μας είναι αυτή της διαφάνειας. Δηλαδή να γνωρίζουμε εκ των προτέρων πού θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα. Και από αυτήν την άποψη θα πρέπει τα κράτη-μέλη εκ των προτέρων να ενημερώνουν για το πώς θα χρησιμοποιήσουν τα διάφορα κονδύλια. Και αν δεν χρησιμοποιούνται όλα αυτά τα κονδύλια στις μεταφορές από ορισμένα κράτη-μέλη, θα πρέπει να το διευκρινίζουν. Το τμήμα των κονδυλίων που δεν θα επανεπενδυθεί στις μεταφορές, πού θα πάει. Θα πρέπει αυτό να καθορίζεται με σαφήνεια από τα κράτη-μέλη. Διαφάνεια λοιπόν. Και το θέμα του εξυγχρονισμού των οχημάτων. Με βάση τις προτάσεις του Κοινοβουλίου της πρώτης ανάγνωσης, το Συμβούλιο σκέφτηκε και τη δυνατότητα της ε, θέσπισης ενός φόρου για, τις, ε, για την ρήπαση από τις αεροπορικές μεταφορές. Επίσης, ε, το θέμα των κονδυλίων αερο 5 και 6. Μιλήσαμε και για την τετραετή προθεσμία για τα ευρώ 6, δηλαδή 5, τέλη του 2017. Στη δική μου πάντως έκθεση εγώ παρέτεινα κατά ένα έτος αυτή την προθεσμία, γιατί προτίμησα ένα περιθώριο λιγμών. Δηλαδή, θα ήθελα το Συμβούλιο να δεχθεί την δική μας πρόταση, τη δυνατότητα, δηλαδή για τα πιο ρηπογόνα οχήματα, να συνδυάσουμε την, το τέλος των υποδομών με το markup, όπως το λέμε, και που ήδη επιτρέπεται για τις ορεινές περιοχές. Θέλουμε λοιπόν ένα συνδυασμό αυτών των μεθόδων για τα οχήματα ευρώ 0, 1, 2 και 3. Όπως είπα, θα μπορούσα να δεχτώ και την τετραετία, την τετραετή προθεσμία, αρκεί να συμφωνήσει το Συμβούλιο με τη δική μας γενική προσέγγιση. Επίσης, καλό θα ήταν υπόψη διαφορά μεταξύ των πιο ρηπογόνων ε, οχημάτων και των ε, εξυγχρονισμένων με στόχο τον όσο και μεγαλύτερο εξυγχρονισμό του, των οχημάτων. Σε ό,τι αφορά την χωρητικότητα, είπαμε ότι θα πρέπει η πρόταση αυτή να ισχύει για τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων. Αυτό προτείνει η οδηγία από το 2012. Το Συμβούλιο πάντως είναι κάπως πιο γενικό και αόριστο στην περίπτωση αυτή και ε, εξασφαλίζει μεγαλύτερο περιθώριο λιγμών για τα κράτη-μέλη εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να προβλέπετε με σαφήνεια στο νομοθετικό κείμενο τι επιτρέπεται και τι όχι και ο μέσος όρος θα πρέπει να είναι 3,5 τόνοι. Σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις θα μπορούσαμε να ξεκινάμε από τους 12, αλλά θα πρέπει να εξηγούμε με σαφήνεια για ποιες ε, προϋποθέσεις πρόκειται και για ποιες συνθήκες. Επίση, τι μέλη γενέστε. Η νομοθετική αυτή πράξη φυσικά δεν θα είναι τέλεια από την αρχή. Θα πρέπει να προβλέψουμε κάποιο μικρό χρόνο για να λάβει χώρα και μια αλλαγή της νοοτροπίας και επίσης για να κερδίσουμε και την κοινή γνώμη. Ούτε με την έγκριση της οδηγίας αυτής ολοκληρώνεται το έργο, γιατί ήδη από την εφαρμογή θα πρέπει να εξετάσουμε και το θέμα της αναθεώρησης και το θέμα της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής αυτής της οδηγίας, για να καλύψουμε και άλλους τύπους οχημάτων και άλλο είδος εξωτερικού κόστους και ούτε καθεξής έχω επίγνωση του γεγονότος ότι για ορισμένες ε, πολιτικές ομάδες ορισμένα τμήματα της πρότασης είτε είναι πολύ φιλόδοξα είτε είναι άτολμα. Πάντως ε, επιμένω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να καταλήξουμε σε κοινή θέση ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να βρούμε μια ρεαλιστική ισορροπία που ταυτόχρονα θα προβλέπει και θα αφήνει και ένα περιθώριο λιγμών και θα κρατήσουμε και κάποια διαπραγματευτικά ατού, ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τη θέση μας όσο γίνεται απέναντι στο Συμβούλιο. Αυτά κύριε Πρόεδρε και ελπίζω οι συνάδελφοι να υποστηρίξουν την προσέγγιση μου. Επίσης, θα ήθελα στις θέσεις μας να είμαστε πολύ ακριβείς και να περιοριστούμε στον αριθμό των τροπολογιών. Νομίζω ότι είναι μία από τις εκθέσεις όπου Φυσικά δεν μπορούν να μείνουν όλοι ικανοποιημένοι και συνέχεια. Ούτε ο Σολομώντας δεν θα μπορούσε. Μόνο, μόνο με τη σοφία του Σολομώντα θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε ικανοποιητική για όλους η λύση. Έχουμε Word McCall, Sterks, Lichtenbergen και Ζήλε από τις ομάδες που είναι οι σκιώδεις ηγητέ. Γκρός, Ρικάουντε, Γκράντε Πασκάλ, Καντσιάν. Στον κατάλογο άλλο κανείς. Φιντάντσα. Ράμε. Yeah, uh, Mr. Durant, Mr. Yeah, Mr. Lightfried and Mr. Van Dalen. Is that it? Let me go through the list again. Ξαναδιαβάζω το κατάλογο ομιλητών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 Το πρόβλημα είναι, κάποια στιγμή θα το μάθω, αλλά θα περάσουν κάποια χρόνια. Ίσως μέχρι το 2014. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Βόρτμαν Κόλ, εκ μέρους του ΕΛΚ. Τέσσερα λεπτά για τους και ηγητές, θα έλεγα και τρία λεπτά για τους υπόλοιπους ομιλητές. Eh, eh, eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συγητή για τη δουλειά που ήδη έχει κάνει. Και αντικατοπτρίζεται η ανταλλαγή απόψεων στην έκθεση. Έγινε συνεργασία στενή τις τελευταίες εβδομάδες και στην ομάδα 2 θεωρούμε ότι πετύχαμε πρόοδο και αυτό αντικατοπτρίζεται σε κάποιο βαθμό στο σχέδιο έκθεσης. Ίσως θα άξιζε τον κόπο εκ μέρους του ΕΛΚ να επενθυμίσουμε ποιες είναι οι προτεραιότητές μας. Πρώτα απ' όλα, να τονίσω το τέλος συμφορήσεως ότι κινείται όσον αφορά αυτό το θέμα το Συμβούλιο προς σωστή κατεύθυνση. Θα θέλαμε περαιτέρω διευκρινήσεις όμως όσον αφορά τις ημερομηνίε πιο συγκεκριμένα. Αναφερόμαστε σε διαφορεοποίηση των τελών. Η τελική μας όμως τοποθέτηση πρέπει να είναι ουδέτερη και πρέπει να υπογραμμιστεί η ανάγκη να εφαρμοστεί σωστά το σύστημα στους δρόμους να αποθαρρύνουμε θέλουμε τα οχήματα να κινούνται την ώρα εχμής. Να βρίσκουν άλλη διαδρομή, να μην από συγκεκριμένε διαδρομέ όπου δημιουργείται συμφόρηση. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα. Θέλουμε περαιτέρω συζητήσει με το Συμβούλιο πάνω σε αυτό. Τις χρονικές περιόδους, τα διάφορα ποσοστά. Αν πάρετε το ποσοστό των 175% μαζί με τα άλλα κριτήρια βλέπουμε ότι είναι σημαντικά στοιχεία. Πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των ορών εχμής και των άλλων ορών. Κάτι άλλο σημαντικό για μας είναι η προσημείωση διαφόρων ποσών. Μπορώ να είμαι σύντομη, διότι ο εισηγητής κινείται προς σωστή κατεύθυνση. ότι πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τη φαιά ζώνη. Η φαιά ζώνη ας είναι όσο το δυνατόν πιο ανοιχτόχρωμη, ας το θέσουμε έτσι. Σας και αγράφησα λοιπόν τη θέση της ομάδας μου. Άλλο σημαντικό στοιχείο για μας, για την ομάδα μας, είναι η διαλειτουργικότητα. Υιοθετήσαμε σχετικά νομοθετήματα. να μπορεί να ταξιδεύει κανείς όλη την Ευρώπη με μια και μοναδική ευρωβινιέτα, αλλά εξακολουθούμε να βλέπουμε διαφορετικές βινιέτες για την ώρα, 6-7 ειδών στο παρμπρίζ των αυτοκινήτων. Θέλουμε τελικά να κάνουμε ό,τι γίνεται τόσο ώστε να εφαρμοστεί σωστά η νομοθεσία. Αυτές ήταν οι προτεραιότητες που είχαμε και έχουμε. Τώρα, όσον αφορά όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για διάφορα εκκρεμή ζητήματα, νομίζω ότι ακολουθούμε τη σωστή κατεύθυνση και θα μπορούν να αυξηθούν τα ποσοστά, αν χρειαστεί κάτι τέτοιο, να, να εισπράττονται τέλη από παράλληλους δρόμους, αλλά θα θεωρείται ανταγωνιστική διαδρομή. Αυτό είναι κάτι που θα συζητήσουμε το Συμβούλιο. Όσον αφορά την ανανέωση του στόλου των οχημάτων, αυτό είναι κάτι που αναφέρθηκε. Το συζητήσαμε εκτενώς το θέμα με το Συμβούλιο. Λέτε εσείς ας κρατήσουμε τα τέσσερα χρόνια, αλλά ας δούμε ποιε είναι οι κατηγορίε των οχημάτων που θα πρέπει να επιβαρυνθούν περισσότερο. Στις ζώνες 1, 2, 3, εκεί ίσως να απαιτείται ένα συμβιβασμό με το Συμβούλιο, διότι υπάρχουν αρκετές αντιστάσεις, δεν υπάρχει ομοφωνία στον αφορά το θέμα, για την ώρα θεωρούμε ότι όσον αφορά τις διάφορες κατηγορίες των οχημάτων είναι σωστή η θέση και μπορούμε να καταλήξουμε σε καλό συμβιβασμό με το Συμβούλιο. Αυτά λοιπόν. Νομίζω ότι αναφέρθηκα στα βασικά σημεία τα οποία αφορούν την ομάδα μου. Η προσέγγιση της Ουγγρικής Προεδρίας είναι επικοδομητική και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να βρούμε μια λύση. Κάποιες τροπολογίες θα υποβληθούν από την ομάδα μου που θα διευκρινίζουν τις διάφορες θέσεις που σας ανέφερα εδώ, κατάθεση τροπολογιών είναι δημοκρατικό μας δικαίωμα και επιφυλασσόμεθα να υποβάλουμε τροπολογίες. Είμαστε επικοδομητικοί. Ο κύριος Τέρξ από την ομάδα Άλτα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα... καταρχήν και εγώ να ευχαριστήσω το ΣΑΙΔ για την καταπληκτική δουλειά που έκανε μέχρι τώρα και που θα συνεχίσει και στο μέλλον γιατί δεν ολοκληρώνεται εδώ το θέμα αυτό. Η κυρία Βόρτμαν Κόλ ασχολήθηκε με πολύ σημαντικά θέματα και ανέφερε ζητήματα που μας ενδιαφέρουν όλους. Το πεδίο εφαρμογή. Να ξεκινήσουμε με τους 3,5 τόνους. Και ευελπιστούμε ότι θα δεχτεί αυτή την πρόταση το Συμβούλιο και θα περιορίσει τις εξαιρέσεις. Ο ξεχρονισμός ε, του στόλου των οχημάτων. Σωστή είναι η κατεύθυνση. Θα δούμε τι θα γίνει με τη διαφοροποίηση των ποσοστών των συντελεστών. Πάντως το γεγονό ότι υπάρχουν είναι πολύ σημαντικό, γιατί μιλούμε 175% το, ή το 200% δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Σε ό,τι αφορά τι ώρε ε, και εκεί μπορούμε να καταλήξουμε συμβαστική λύση και συμφωνώ με την πρόταση του εισηγητού. Σε ό,τι αφορά τον προορισμό των ε, κονδυλίων, αυτό το θέμα για μένα είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αν δεν συμφωνήσουμε με τα κράτη-μέλη ώστε τα έσοδα αυτών των τελών να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των υποδομών και του συστήματος των μεταφορών, να επενδυθούν δηλαδή στις μεταφορές, τότε κάπου θα έχουμε κάνει λάθος. Αυτό το γνωρίζει θαυμάσιο εισηγητή και νομίζω ότι και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε τελικά σε συμφωνία με το Συμβούλιο για την επανεπένδυση στις μεταφορές. Μία άλλη τροπολογία, γιατί βρίσκω Καταρχήν βρισκόμαστε στην αρχή μιας ε, ευρείας συζήτησης. Οπότε καλό θα ήταν να καθορίσουμε διάφορες αρχές ό,τι αφορά το εξωτερικό κόστος, αν θα γίνει καταλογισμός τους κάπου ή όχι. Πρόκειται για το, την πρώτη νομοθετική πράξη ε, που έχουμε για τον τομέα αυτό και θα χρησιμοποιηθεί ως σημείο μεταφοράς, ε, ως σημείο αναφοράς, συγγνώμη, και για τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς. Πρόκειται για μια νομοθετική ρύθμιση που θα αναλυθεί διεξοδικά την επόμενη δεκαετία, αλλά τα θεμέλια θα μπουν από τώρα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να καθορίσουμε τις γενικές αρχές πέραν των λεπτομεριών και να δούμε πώς ε, θα μπορέσουμε να τις εφαρμόσουμε στην πράξη. Πάντως ε, το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να θεσπίσουμε κάποιες αρχές. Αυτό είναι σημαντικό για το μέλλον γιατί θα χρησιμοποιηθούν αυτές ως σημείο αναφοράς. Το Συμβούλιο είναι υπερβολικά περιοριστικό. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο ευρύ στις ε, προσεγγίσεις μας και συμφωνώ με τον εισηγητή ότι καλό θα ήταν στην Επιτροπή μας να ακολουθήσουμε μια γραμμή συνενετική την οποία θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε όλοι και καλό θα ήταν ο εισηγητής να έχει και άτυπες επαφές με το Συμβούλιο για να κάνει μια βολιδοσκόπηση και να μας πει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως καταφέραμε μέχρι στιγμής να καταλήξουμε σε μια συνενετική θέση που ελπίζουμε ότι θα γίνει δεκτή από το Συμβούλιο. Και εκεί έγινε το κίνδυνος. Κάποιες χώρες του Συμβουλίου να μην συμφωνήσουν με αυτές τις αρχές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό από πολιτική άποψη. Αυτό όμως είναι, αυτός είναι ένας κίνδυνος που ελοχεύει και αυτή τη στιγμή δεν, θα το... δεν χρειάζεται να μας απασχολεί, θα το δούμε αργότερα στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ κυρία Λίχτεμπεργκερ για τους πράσινους. Yeah. Ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε. Αν παραμείνω στην ίδια εικόνα της ε, συναδέλφου Λοτμαν δεν προχωρήσαμε σε λιγότερο φαιά ουσία προς το άσπρο, τουλαντίον πολύ σκούρο γκρι το βλέπω. Αυξάνονται τα κασάρια. Θα πρέπει να ξέρουμε τι συζητάμε αυτή τη στιγμή σε αυτό τον φάκελο όσον αφορά την ανανέωση του στόλου, όσον αφορά την προστασία των κατοικών στην, ε, στα στο περίγυρο των οδών αυτών, τίποτα δεν κάνουμε. Περιθωριακά τέλο πάντων κάτι κάνουμε ελάχιστο. Το μόνο που πετύχαινουμε είναι να αναγνωριστεί η αρχή ότι υπάρχει δηλαδή ένα εξωτερικό κόστος. Τίποτα άλλο. Αλλά το πρόβλημα είναι το εξή. Οι αρχές από μόνες τους δεν ωφελούν όταν αυξάνεται ο ρυθμός χρήσης αυτών των ε, των οδών και όταν θέλουμε να προστατεύσουμε καλύτερα το κλίμα. Κάποια στιγμή δηλαδή θα πρέπει να περάσουμε σε μια πρακτική εφαρμογή, αλλιώς ε, κινδυνεύει η αξιοπιστία μας. Όσον αφορά το λεγόμενο earmarking, τον καθορισμό δηλαδή κάποιων κονδυλίων για συγκεκριμένα θέματα που για σας είναι τόσο σημαντικό. Μου φαίνεται κάπω ε, εικονική η μάχη αυτή, γιατί όλες οι χώρες που εισπράττουν από την Ευρωβινέτα θα προβλέψουν στον συγκεκριμένο τομέα λιγότερους πόρους στους προπολογισμούς τους. Λόγω και της δημοσιονομικής κρίσης που ζούμε αυτή τη στιγμή. Δεν θα αλλάξουν λοιπόν πολλά πράγματα. Αν υπάρχει λίγο έσοδο, ε, θα πρέπει να προβλεφθεί κάτι παραπάνω στον προλογισμό του εν Αυτό είναι μάλλον συμβολικής αξίας και όχι πρακτικής και ουσιαστικής. Κάτε με, ναι. δύο σημεία είναι πάρα πολύ ουσιαστικά για να πετύχουμε κάπου ενδεχομένως κάποιο αποτέλεσμα. Πρόκειται για την προσθήκη αυτή του λεγόμενου markup. Θα πρέπει να γίνει από το 1 στο 3. Από το 1 στο 3 όμως δεν θα έχει καμία επίδραση. Γιατί η τάξεις αυτές των ε, φορτηγών δεν έχουν πάρα πολύ σημαντική επίπτωση στις ε, μεταφορές μεγάλων αποστάσεων. Ας πούμε τέσσερα επιπλέον για να έχουμε ένα μικρό κίνητρο για τη βελτίωση των στόλων. Ένα ελάχιστο θα ήταν αυτό, μια ελάχιστη πρόταση. Το δεύτερο, η διατύπωση όσον αφορά τους 12 τόνους και τους 3,5 τόνους θα πρέπει να είναι πάρα πολύ ακριβείς ε, για να είναι σαφές ότι πρόκειται για ένα περιορισμό. Αλλιώς, η ε, τελευταία λύση θα επιδεινώσουμε την κατάσταση. Το ότι αξιολογείται επίσης ο θόρυβος μόνο τη νύχτα δεν μου φαίνεται σωστό, ούτε και ιατρικά είναι σωστό. Γιατί βέβαια ε, η η χορύπανση επιδεινώνεται εάν ε, επιδρά 24, 36 ή 48 ώρες. Δηλαδή η μείωση αυτή των πολλαπλασιαστών για μένα είναι πάρα πολύ ενοχλητική. Στις τροπολογίες ε, του Ελκατράου δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα αρνητικό εκτός από το θέμα αυτό της θέσης ισχύει. με τα markups και το εξωτερικό κόστος. Πολλές από αυτές τις τροπολογίες θα μπορούσα κάλλιστα να τις ε, υποστηρίξω. Θα πρέπει για δύο-τρεις να δούμε ποια θα είναι η τελική διατύπωση. Αλλά δεν υπάρχει πια καμία φιλοδοξία. Αναρωτιέμαι λοιπόν γιατί το ΕΛΚ προσπαθεί ακόμα να αποδυναμώσει περισσότερο. Υπάρχει μάλιστα και μια δία που λέει ίσως υπάρχει εξωτερικό κόστος. Αυτό περιμένω να δω τουλάχιστον. Γιατί αυτό σήμερα δεν θέλουν τίποτα. Περιμένω δηλαδή να ακούσω να διαφεσβητείτε ε, η λήψη υπόψη του εξωτερικού κόστου. Στην πραγματικότητα δεν βλέπω να υπάρχει καμιά αλλαγή και δυστυχώς ομολογώ ότι να το εξηγήσουμε αυτό στους πολίτες που κατοικούν εκεί στις, ε, σε αυτές τις ε, κύριες οδούς ε, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία, αλλά η, ε, μια αρχή δεν θα βοηθήσει κανέναν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Σίλοφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ελκαντράου για τη δουλειά που έκανε Έγινε καλή προσπάθεια συντονισμού και πρέπει να συμφωνήσουμε επί των στόχων μας. Σαν κοινοβούλιο για να έχουμε θέση στις διαπραγματεύσεις του το Συμβούλιο. Νομίζω ότι γενικά όμως σημειώνουμε μια πρόοδο. Πρέπει να συμβιβαστούμε τελικά με το Συμβούλιο. Η ομάδα μας έχει ε, διάφορες προτάσεις. Η μία αφορά τον μέγιστο αριθμό ωρών να είναι 8 ώρες το όριο, ενώ το Συμβούλιο λέει 5. Πρέπει να προχωρήσουμε, να κάνουμε ένα βήμα πιο πέρα και να βρούμε μια λύση ανάμεσα στις 5 ώρες και στις 8 ώρες. Τώρα, μέγιστη διαφοροποίηση μπορεί να είναι 200% πάνω το μέσο όρο ή 175% όπως προτείνει το Συμβούλιο. Μπορούμε να βρούμε μια μέση λύση, πιστεύω. Θα αποτελέσει και πολιτική χειρονομία το να συμβιβαστούμε με το Συμβούλιο. Και μετά μπορούμε να συγκεντρωθούμε επί άλλων θέσεων. Και πρέπει να περασπιστούμε στεναρά μια άλλη θέση του Κοινοβουλίου για το θέμα του Μάρκαπ, το περίφημο. Όσον αφορά την ανανέωση του στόλου των οχημάτων, θεωρήσαμε ότι οι θέσεις του Συμβουλίου ήταν καλύτερη. Τα διάφορα κράτη-μέλη έχουν ανταγωνιζόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα είναι δύσκολο για αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο μέλλον η όλη κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουν και δεν θα τους βοηθούσε εάν δεν ληφθούν τα σωστά μέτρα, κυρίως στις επιχειρήσεις που έχουν μικρό μερίδιο της αγοράς στην εσωτερική αγορά της Ευρώπης. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Ένα υγιές περιβάλλον. Αυτή πρέπει να είναι πρώτη στη μνά μας. Πάνω σε αυτό λοιπόν Πιστεύω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε με τον εισηγητή για να καταλήξουμε σε κάποιες συμβαστικέ λύσεις για να διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο. Κεντρική ιδέα ποια είναι ότι το σύστημα έβρεση θα πρέπει να είναι το σωστό για να δημιουργεί τη σωστή ατμόσφαιρα της επιχειρήσης. Όσον αφορά τη μόλιση του περιβάλλοντος, ο ρηπαίνων θα πρέπει να πληρώνει. Αν τα τέλη είναι υπερβολικά, τελικά θα, αποθαρρυνθούν θα αποθαρρυνθεί ο κόσμος και θα βγαίνει καν με τα αυτοκίνητα στο δρόμο. Και πρέπει να υπάρχει μια γενικότερη κάλυψη. Ευχαριστώ κύριε Ζήλε. Πάμε στα μέλη. Γενικώ, σύντομα τρία λεπτά για να έχουμε χρόνο να ακούσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κ. Γκρό λοιπόν ξεκινάει το τριλεπτό του. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Εργάστηκε πολύ καλά και δεν σας αποκλείω ότι εμείς στο ΕΛΚ δεν θα βρούμε εύκολα μια κοινή θέση. Γιατί ειλικρινά έχουμε να κάνουμε με συναδέλφους που έρχονται από χώρες που πληρώνουν πολύ και έχουν λίγα έσοδα, ενώ άλλοι θα έχουν πολλά έσοδα και θα πληρώνουν κάτι λιγότερο ίσως. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που υπάρχει και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε. Και εμείς γι' αυτό, ΣΕΛΚ, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μια μέση εδώ όχι μόνο προς όφελος των δικών μου συναδέλφων, αλλά και του ίδιου του θέματος. Δεύτερον, η συνεργοποίηση του κόστους. Αυτό είναι μια αρχή που μπορούμε να δεχτούμε. Θέλουμε όμως να τονίσουμε ότι αυτή η εξέταση θα πρέπει να γίνει σε όλες τις μορφές μεταφορών, όχι μόνο σε οδικές μεταφορές και όχι μόνο στα φορτηγά. Τα φορτηγά είναι ε, ο κύριος στόχος όταν μιλάμε για εσωτερικοποίηση, γιατί πολλοί δεν τα αγαπούν, αλλά θα πρέπει νομίζω στο μέλλον να ε, εξετάσουμε και τους άλλους τομείς και χώρες που προσπάθησαν να συμπεριλάβουν και τα ιδιωτικά οχήματα ξέρουν πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπίσει κανένας το πρόβλημα στη ρίζα του. Ξέρουμε επίσης ότι σήμερα είναι δύσκολη η εναρμόνιση γιατί εδώ η εσωτερικοποίηση του κόστου η Ευρωβινιέτα δεν είναι υποχρεωτική. Δεν καταφέραμε να το καταστήσουμε αυτό υποχρεωτικό. Ξέρουμε ότι εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσπαθήσουμε να υποστηρίξουμε όλα αυτά που λέγονται μέσα στα πλαίσια της εναρμόνισης. Ξέρουμε, 120 χώρες, στη, ε, συγγνώμη, στην Ευρώπη έχουν εισαγάγει μέτρα περιορισμού των εκπομπών μέσα στην αστική περιοχή και πρέπει να φροντίζουμε να μην διαφοροποιηθούν τόσο πολύ οι νόμοι από χώρα σε χώρα. Θα πρέπει να φροντίσουμε εδώ στο Κοινοβούλιο να μην έχουμε μόνο τη γενική συζήτηση του εσωτερικοποίησης του κόστους, αλλά να προωθήσουμε και την εναρμόνιση. Και γι' αυτό μου φαίνεται ότι το λεγόμενο ERMAC είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι κεντρικό θέμα. Επίσης, η διαλειτουργικότητα το ίδιο και η εναρμόνιση ε, επίσης και για το υπόλοιπο της συζήτηση δεν θα πρέπει να... Ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε μάλλον να προχωρήσουμε με το Συμβούλιο όσο μπορούμε, γιατί ξέρουμε ότι με το Συμβούλιο υπάρχουν προβλήματα, γιατί το 50% των χωρών δεν θέλουν ευρωβινιάτα. Ας είμαστε λοιπόν λογικοί και α προσπαθήσουμε να πετύχουμε τι καλύτερε δυνατέ συμβαστικέ λύσεις. Το να είμαστε υπερβολικοί στις μα μας δεν νομίζω θα μας οδηγήσει πουθενά. Καλύτερα να σκαλώσει ο Ευχαριστώ. Ο κύριο Λάιτφριτ, τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Αυτό που θα σας πω τώρα, να μην το εκλάβετε σαν επίκριση του εισηγητή που εργάζεται σκληρά οπωσδήποτε. Ομολογώ όμως ότι δεν έχω ικανοποιηθεί. Ήδη δεν είχα ικανοποιηθεί όταν αποφασίσαμε τα θέματα αυτά στην πρώτη ανάγνωση. Το είπε ο κύριος Κρός. Ε, θα πρέπει να υπάρχουν ελάχιστα διόδια για, τις, για τα ευρωπαϊκά ε, δίκτυα είχαμε πει στο παρελθόν. Δεν το πετύχαμε αυτό. Δεν πετύχουμε επίσης στους εξωτερικούς παράγοντες να συμπεριλάβουμε τις ε, εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε ότι οι βαριές οδικές μεταφορές που μου το περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα δεν εντάσσονται μέσα στους κανονισμούς και το διοξείδιο του άνθρακα. Αυτά είναι η στιγμή που πραγματικά με αφήνουν ανικανοποιητό. Δεν είμαι καθόλου ευτυχής για την ε, απόφαση που ελήφθη τότε. Και μετά την απόφαση του Συμβουλίου είμαι ακόμα λιγότερο ικανοποιημένο. Είναι για μένα τελείως ακατανόητο. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε συμπληρωματικό κόστος ε, που να συνδυάζει το κόστος για τις ευαίσθητες ε, περιφέρειες. Γιατί όσον αφορά την χορύπανση έχουμε μειώσει τα αριθμητικά στοιχεία του Συμβουλίου τόσο πολύ που δεν υπάρχει πια καμία κύρωση. Και ακριβώς στους ε, περιοχές που δεν κατοικούνται όπως τις ε, ορεινές κοιλάδες δεν υπάρχει καμία επιβολή ε, μάλλον δεν λαμβάνεται κανένα εξωτερικό κόστος υπόψη για την ηχορύβανση τι να κάνουμε. Υπάρχει αυτή η θέση που υπάρχει, πρέπει να προσπαθήσουμε να τη βελτιώσουμε. Και δεν ξέρω, θα πάμε στι διαπραγματεύσει με λίγα ή με πολλά. Εγώ είμαι μεταξύ εκείνων που λέει ότι όσο πιο πολλά έχει κανένα μπαίνοντα σε μια διαπραγμάτευση, τόσο πιο πολλά έχει και βγαίνοντα από αυτή. Και θεωρώ ότι αυτή η Επιτροπή, αυτό το σώμα θα ήταν σωστό να ο, καταγράψει αυτά που θεωρούμε εμεί σωστά χωρί να λάβει υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου. Και θα δούμε μετά ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Καταρχήν, η συμπερίληψη του εξωτερικού κόστου είναι ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση. Αλλά το βήμα αυτό δεν είναι βήμα, αλλά τι να σας πω, είναι ούτε βηματάκι καν, δεν θα έχουμε τελικά κανένα αποτέλεσμα. Και θα αναγκαστούμε να καταψηφίσουμε και αυτού του δικαιώματο επιφυλάσσουμε κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Λάιτφριτ. Για τρία λεπτά η κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τον κύριο Ραχαντράουι για το έργο του και την προσπάθειά του. Αλλά και εγώ έχω κάποιε δυσκολίε όπω είπε και η συνάδελφο. Θα πρέπει να προβούμε σε μια στρατηγική επιλογή. Πού θα βάλουμε τον πύχη. Πολύ ψηλά ή θα αρχίσουμε από την αρχή να αποδυναμώνουμε το κείμενο. Επίσης ε, και το θέμα της Λευκής ε, Βίβλου. Θα πρέπει να είμαστε αρκετά φιλόδοξοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε ό,τι αφορά την επανεπένδυση στον τομέα των μεταφορών, φυσικά είναι καλή ιδέα ή μάλλον δεν είναι κακή ιδέα της επανεπένδυσης των εσόδων αυτών, αλλά δεν είναι ικανοποιητικά αυτά τα κριτήρια σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα που θα έχουν τα κράτη-μέλη, την υποχρέωση που θα φέρουν να επενδύσουν σε χρήσιμα θέματα για τις μεταφορές. Στα κριτήρια της τροπολογίας 18 φοβούμε ότι ε, με τις επενδύσεις αυτές τα κράτη-μέλη θα μειώσουν τον προϋπολογισμό τους ε, για τις μεταφορές ε, γιατί με την Ευρωβινιέτα τελικά δεν θα γίνει η εσωτερήκευση του κόσμου, απλώς θα ελαφρυνθεί ο προϋπολογισμός των κρατών μελών για τις μεταφορές. Δηλαδή τα κράτη-μέλη θα κάνουν σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι ο στόχος της Ευρωβινιέτας σε ό,τι αφορά τις ώρες της αιχμής. Τελικά με τα συνολικά αποτελέσματα θα είναι πολύ πιο φθηνές οι οδικές μεταφορές για όλους. Γιατί είναι αρνητικό το κόστος συμφόρησης στι ε, μία ώρες εχμής γιατί έχουμε ψηλότερη εισφορά στις ώρες αιχμής και στις ώρες αιχμής τελικά θα πληρώσουμε λίγο περισσότερο για να ε, κυκλοφορούμε λιγότερο, αλλά θα γλιτώσουμε τη, τα ποτηλιαρίσματα. ποιο είναι τελικά το αποτέλεσμα, θα είναι πιο φθηνές οι οδικές μεταφορές. Αυτός είναι ο στόχος της ε, εσωτερήκευσης. Και, αυτό που είπε η κυρία Λιχτεμπέργκερ. Και εγώ με, και εγώ ενδιαφέρομαι για το θέμα του, του κλάδου και να στηρίξουμε τους μεταφορείς γιατί αντιμετωπίζει δυσκολίες αλλά θα πρέπει να στείλουμε και ένα ηχηρό μήνυμα. Τι θέλουμε. Δεν είμαστε κατά των οδικών μεταφορών αλλά θέλουμε να ενθαρρύνουμε έναν κλάδο και να δώσουμε τα μηνύματα για το τι περιμένουμε από τον κλάδο αυτό. Θέλουμε διαλειτουργικότητα και συνδυασμένες μεταφορές. Δεν θέλουμε να ενισχύσουμε ανεφόρα το τομέα, να το ενθαρρύνουμε και να έχουμε και πιο ε, οικολογικέ μεταφορέ. Προτιμώ να βάλουμε τον πύχη ψηλά στην αρχή, ακόμη και αν αυτό θα γίνει με το τίμημα τη αντιπαράθεση ε, προ το Συμβούλιο, αλλά νομίζω ότι έχει νόημα να είμαστε πολύ φιλόδοξοι, ειδικά στην αρχή. Τρία λεπτά ο κύριος Βαντάλεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ και μία δεκαετία ασχολούμαστε με το θέμα αυτό και φαίνεται ότι πλησιάζουμε στην κατάληξη και νομίζω ότι καλό θα είναι να δείξουμε μία υπευθυνότητα και να αξιοποιήσουμε τα μέχρι τώρα αποτελέσματα και επιτεύγματα. Βέβαια, σίγουρα κάποιες ε, πολιτικές ομάδες είναι απογοητευμένε και θα προτιμούσαν κάποια πιο φιλόδοξη εξέλιξη, αλλά νομίζω ότι ποτέ δεν ήμασταν τόσο κοντά σε αίσιο πέρα σε ό,τι αφορά ε, την ε, εξωτερήκευση, για παράδειγμα, του κόστους. Σε ό,τι αφορά τα σχόλια του εισηγητή, για τη διαλειτουργικότητα καταρχήν. Ο εισηγητής έχει καταθέσει πολλές τροπολογίες που με βρίσκουν σύμφωνο. Παρ' όλα αυτά όμως στην ε, Ευρώπη έχουμε διαφορετικά συστήματα, διαφορετικές βινιέτες, διαφορετικό σύστημα διοδίων και θα προτιμούσα να έχουμε μια πιο συγκεκριμένη τροπολογία που θα καταθέσουμε ως ομάδα για την διαλειτουργικότητα σε σχέση με τα κείμενα του Συμβουλίου και του εισηγητού που δεν είναι αρκετά φιλόδοξα στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων θα καταθέσω συγκεκριμένη τροπολογία για το θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία Ελκατράουι για την εξαίρεση για το, εξαίρεση για το ευρώ 6 που μιλάει για την τριετία. Δεν καταλαβαίνω. Εμείς μιλούμε για καθαρές ε, οδικές μεταφορές και θέλουμε να ενθαρρύνουμε στην Ευρώπη τη χρήση πιο φιλοπεριβαλλοντικών και πιο καθαρών βαρέων οχημάτων. Οπότε αυτό το στόχο θα πρέπει να έχει και πρόθεσή μας ε, και πρότασή μας για το ευρώ 6, σε αντίθεση με την πρόταση του εισηγητού που μιλάει για εξαίρεση. Μία τέτοια εξαίρεση θα βάλει σε πειρασμό τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν περισσότερο, για περισσότερο χρόνο τα πιο ρηπογόνα οχήματα που είναι τα ευρώ 5. Θα ήθελα να ακούσω τον κόδωνα του κινδύνου λοιπόν ως προς την τροπολογία Ελχαντράουι για τα ευρώ 6. Θα συνεχίσουμε πάντως τις συζητήσεις και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να επομιστούμε τις ευθύνες, να τις ευθύνες μας και να περιορίσουμε στο ελάχιστο τον αριθμό των τροπολογιών. Ευχαριστώ κύριο Ζήκε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς να συγχαρώ τον Σαΐντ για την ευαίσθητη αποστολή του αυτή. Γενικό σχόλιο. Βλέποντας από μακριά το θέμα, θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν πολλά προβλήματα διότι ακολουθούμε βασική αρχή ο, ο ρηπαίνων πληρώνει και εσωτερήκευση του κόστους. Και εν γέννη υπάρχει υποστήριξη. Βλέπουμε ότι το θέμα είναι περιπλοκότατο όμως εκ του συνέγγις και παρακολούθησα με μεγάλο ενδιαφέρον τις περίπλοκες παρουσιάσεις γεμάτες ευαισθησίες και μικροδιαφορές του εισηγητού και των σκιωδών εισηγητών και υπονοούνταν διάφορα πράγματα και δεν λεγόταν ξεκάθαρα. Τα σημεία απόκλησης καλύπτουν περισσότερο τις ομάδες και επηρεάζουν τις τοποθετήσεις. Υποστηρίζω στεναρά τη θέση του συγητού. Τις θέσεις του συγητού που είναι συνετές οι θέσεις, συμβιβαστικές, Ξέρουμε ποια είναι η θέση του Συμβουλίου που είναι πολύ άκαμπτη με μικρά περιθώρια λιγμών. Χρειάζεται μεγάλη συζήτηση για το πώς προς τα που θα κινηθούμε. Είναι θέμα τακτικής και όχι θέμα ουσίας. Θέλουμε το earmarking, την προσημείωση ποσών. Η μεταφορά που ήθελε η κυρία Ντουρό θεωρώ ότι ίσως είναι περίπλοκος σαν προσέγγιση για τις εξαιρέσεις. Ευαίσθητο θέμα. Γιατί να εξαιρέσουμε, μειώσουμε τις εξαιρέσεις του ευρώ 6. Είναι κάτι που μοιράζομαι σαν θέση με το ΣΑΙΔ και να βάλουμε τις κατηγορίες 1, 2, 3 διότι αν έχετε πάρα πολλέ εξαιρέσεις αποδυναμώνεται από το περιεχόμενο την οδηγία. Αν όλα τα βαριά οχήματα πενταετία εξαιρεθούν, μπορούμε να ξαναψηφίσουμε σε μερικά χρόνια το θέμα και να μην το συζητάμε τώρα διαμόρφωση τώρα των τελών, των διοδίων. Εγώ θα ξεπερνούσα το 200%. Είναι το βασικό θέμα το τέλος της συγχώρησης. Και αν θέλουμε μηδενικό τελικό σύνορο, θέλουμε να διαμορφώσουμε και να, την κυκλοφορία και όχι να καταπολεμήσουμε απλώς τη συμφόρηση. Υπερασπίζομαι τον ορισμό του διαδρόμου, του corridor, που θέτει ο ε, εισηγητής και μετά και η ρήτρα του ραντεβού είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί το λέμε ότι γιατί περίζουμε σε μερικά χρόνια να βελτιωθεί η κατάσταση και να έχουμε καλύτερη, να μπορούμε να βρούμε καλύτερες λύσεις. Τέλος, να επενθυμίσω σε εκείνους που δεν υποστήριζαν ένθερμα αυτού του είδους τα κείμενα ότι αν είναι αδύναμη η ευρωπαϊκή θέση, ενθαρρύνονται κάποιες χώρες δυνάμει επικουρικότητας να πάρουν πιο στεναρή θέση. Και τελικά δεν εφαρμοστούν σωστά τα μέτρα. Εάν δεν υπάρχει περιεχόμενο σε διατάγματα ευρωπαϊκά, θα υπάρχουν χώρες που θα εφαρμόζουν τα δικά τους τέλη, τα δικά τους διόδια με πολύ πιο σκληρό τρόπο από ό,τι θα έκαναν αν υπήρχε ευρωπαϊκό πλαίσιο, ευρωπαϊκή νομοθεσία πιο καλά διαθρωμένη. Τι θέλω να πω λοιπόν, προσοχή, υπάρχει ένας κίνδυνος και για εκείνους που είναι κατά τέτοιου είδους νομοθεσίας. Τι θα γίνει, να εξαφαλιστεί η Ευρωβινιέτα υπέρ εθνικών μέτρων που θα είναι ακόμα αυστηρότερα. Αυτά έχω να πω. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ντεγκράντες Πασκάλ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι κανένα δεν θα πρέπει να σκανδαλίζεται, γιατί για το παλιό θέμα της Ευρωβινιέτας, η σύμπτωση ευμενών θετικών κριτηρίων ή η σύγκληση επιχειρημάτων διαφωνίας δεν θα πρέπει να εκπορεύονται από ιδεολογικούς λόγους, αλλά από ζωτικά ή εύλογα εθνικά συμφέροντα. Στα θέματα της Ευρωβινιέτας υπάρχουν ε, πολλοί λόγοι για τις ε, πιο περιφερειακές χώρες που είναι κατά, γιατί θεωρούμε ότι βλέπτονται τα εύλογα μας ε, και ένομα μας συμφέροντα. Γιατί έτσι, σε μια ήδη έφεραυστη οικονομική συγκυρία, θα έρθουμε σε ακόμη χειρότερη κατάσταση και δεν το κάνουμε αυτό από ιδιοτροπία, αλλά φαίνεται να μιλούμε για την τιμή της του χαβιάρι, ενώ σε ορισμένες χώρες ε, με το μισθό τους οι άνθρωποι δεν μπορούν καν ε, να, πληρώσουν τα, τα στοιχειώδη, τις στοιχειώδεις βιοποριστικές τους ανάγκες. Περίπου 57% του εξωτερικού εμπορίου γίνεται στις, με οδικές μεταφορές στην Ισπανία. Και μάλιστα οι προορισμοί ε, των ισπανικών εξαγωγών είναι η Γαλλία και η Γερμανία. 30% των εξαγωγών πάνε στη Γαλλία και το 38% των εισαγωγών προέρχεται από τη Γαλλία και μάλιστα από τις οδικές μεταφορές. Οπότε με τον υπολογισμό αυτό θα είχαμε εκατομμύρια ευρώ επιπλέον συμπληρωματικό κόστος ε, για τις ε, ισπανικές οδικές μεταφορές, κάτι που θα οδηγήσει σε απώλεια της ανταγωνιστικότητάς μας. Το ίδιο και με τη Γερμανία. Το συμπληρωματικό κόστος για τον ε, κλάδο θα είναι πάλι ε, πολλά εκατομμύρια ευρώ. Είναι ελάχιστα αυτά τα παραδείγματα που δικαιολογούν όμως τη γνωστή ισπανική θέση. Να προσθέσουμε σε αυτό το γεγονός ότι η βελτίωση της καθημερινής συμφόρηση δεν γίνεται με την ε, επιβάρηση ορισμένων μονοχημάτων. Επίσης, ε, έτσι θα καταλάβετε καλύτερα τη θέση μας. Πάντως, Καταλαβαίνουμε το Συμβούλιο έκανε σημαντικέ προσπάθειε, το ίδιο και ο εισηγητή. και μάλιστα διευκρίνησε ο εισηγητή ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι όχι να απορρίψουμε, αλλά να βελτιώσουμε τη θέση του Συμβουλίου στη δεύτερη ανάγνωση. Θα πρέπει να είμαστε χρήσιμοι και να δείξουμε πνεύμα συνεργασία. Θα μπορούσαμε να πούμε υπέρ του εισηγητού ότι όντω διαφοροποίησε τι θέσει του και πραγματικά ήταν ελαστικό και διαλλακτικό και το αναγνωρίζουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι τροπολογίε του εισηγητού, θα προσπαθήσουμε να είμαστε συνεργάσιμοι και διαλεκτικοί, Σε ό,τι αφορά την ε, επανεπένδυση του κόστους ε, ε, του, των εσόδων από, τα, από το εξωτερικό κόστος, συμφωνούμε με την τροπολογία 18 που μιλάει για την επανεπένδυση των χρημάτων αυτών προκειμένου να βελτιστοποιηθεί το σύστημα των οδικών μεταφορών. Νομίζω ότι βελτιώνεται έτσι η θέση του Συμβουλίου. Πάντως το 15% αυτών των εσόδων θα αφιερωθούν στα διευρωπαϊκά δίκτυα χωρίς να προσδιορίζεται. Δεν είναι δίκαιο αυτό. Σε ό,τι αφορά την διασταυρώμενη χρηματοδότηση θα βλάψει τις οδικές μεταφορές και θα ευνοήσει τους ανταγωνιστές της. Από τη στιγμή που οι οδικές μεταφορές θα πληρώσουν το τίμα, θα πρέπει αυτές να υποφεληθούν και από τι δαπάνε αυτέ, Γιατί μην ξεχνάτε ότι με τι οδικέ μεταφορέ εξασφαλίζουμε το εσωτερικό εμπόριο τη Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά το τέλο για τη μείωση τη συμφόρηση. Συμφωνώ με τη διαμαρτυρία του εισηγητού στην τροπολογία 5, γιατί δίνεται μια χρηματοοικονομική αντιστάθμιση στου χρήστε των, των δρόμων στι στις ε, περιόδους που δεν είναι ώρες εχμής. Επίσης, συμφωνώ με την ε, αύξηση των ωρών εχμής που συνδυάζεται και με τη διαφοροποίηση του τέλους. Κύριε Ισηγητά, θετικές είναι και οι τροπολογίες σας προς τα κράτη-μέλη που θα πρέπει να ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για, για την εφαρμογή της οδηγίας, τροπολογίες 6 και 10. Σε ό,τι αφορά τον καθορισμό του διαδρόμου για την επιβάρηση, και το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνουν ό,τι μπορούν για να καταλήξουν συμφωνία. Ο κύριος Αλκαντράουι κατέθεσε την τροπολογία 6 που μιλάει για την επιβάρηση που θα πρέπει να επιβάλλεται σε εναλλακτικέ διαδρομές. Τελικά ο ο εισηγητής έδειξε ελαστικότητα απέναντι και στη θέση του Συμβούλιο. Αυτά κύριε Πρόεδρε, θα καταθέσουμε και τροπολογίες για να ε, στηρίξουμε τις θέσεις μας. Θα ήθελα να επενέσω τον ε, εισηγητή που πραγματικά κάνει πολύ λεπτεπίλεπτη προσπάθεια και είναι περίπλοκο το έργο του. Αναγνωρίζουμε την προσπάθεια, αλλά μην ξεχνάτε ότι εξαιτία των ε, ένομων και εύλογων ε, εθνικών συμφερόντων είναι λογικό να υπάρχουν και διστάμενες απόψεις πολλές φορές για κάποια σημεία. Τρία λεπτά ο κύριος Καντσάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ, Σαΐτ, και πραγματικά δεν συζηλεύω καθόλου για, την ε, θέση που έχεις, ε, για τη θέση που έχεις ε, με την ιδιότητά σου ως εισηγητής αυτού του ζητήματος που είναι πολύ περίπλοκο. Μιλήσαμε για την ανήψη του πύχη, για την ανάγκη μεγαλύτερης φιλοδοξίας. Για τα θέματα αυτά όμως θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποιες σκέψεις. Τι συμβαίνει εδώ. Πέραν της αρχής ότι ο χρήστη πληρώνει θα πρέπει να προσθεθεί στο ρηπένον πληρώνει είναι αποδεκτή, λογική, αρχή και μας βρίσκει σύμφωνου. Ναι. Και σε ό,τι αφορά το, ε, το επιπλέον τέλος, το συμπληρωματικό τέλος, το συμπληρωματικό, πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι ουδέτερο. Λοιπόν, θα δανέμουμε το κόστος λοιπόν των τελών ώστε να διαφυλάξουμε την αρχή. Αν αντίθετα σήμερα, όπως κάνουμε πέρα από την οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουμε, και εξετάσουμε ιδιαίτερα το θέμα των οδικών μεταφορών και την κατάσταση επικρατεί, εμείς οι πολιτικοί που θα πρέπει να διερευνήσουμε το πώς μπορούμε να θεσπίσουμε νόμους για τις υποδομές, ανανέωση των παλαιών στόλων των οχημάτων, τη διαλειτουργικότητα, για να μην έχουμε συμφορήσεις. Ε, να διαφυλάξουμε και τις διάφορες ε, που έχουν γίνει να φροντίσουμε λοιπόν τελικά να υπάρχει επανεπένδυση για δημόσια έργα, τέτοια περίοδο κρίση που περνάμε, αν θέλουμε να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα, αρκεί να αναβάσουμε απλώς τα τέλη για να τα πληρώσουμε όλα αυτά. Αυτή είναι η ευθύνη μας, έτσι αντιμετωπίζουμε την ευθύνη μας. Δεν είναι αυτή η ευθύνη μας. Η ευθύνη μας ως πολιτική είναι να προβλέψουμε να υπάρξουν υποδομές, να γίνει ανταλλαγή των οχημάτων, να υπάρχει διατροπικότητα, αν θέλετε, διαφόρων μέσων μεταφοράς, πέρα από την κατηγορία που, τη συγκεκριμένη που εξετάζουμε. Δεν πρέπει να είναι πολύ απλουστευμένη η προσέγγιση όσον αφορά την εφαρμογή απλώς μία αύξηση του, του τέλους και μετά το κόστος να εσωτερικεύεται και να προσπαθεί να καλύψει τις δικές μας ελλείψεις. Κατά την άποψή μου δεν είναι αυτή η λογική της πολιτικής. Η πολιτική ασκείται με άλλο τρόπο, ε, με διαφορετική προσέγγιση φορά του με διαφορετικό προγραμματισμό, διότι ο απλός χρήστης θα μας πει θα διαμαρτυρηθεί αν πρέπει να υπομειστεί όλα τα βάρη στους ώμους του για να μπορεί να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό του είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς την απλούστευση που ακολουθούμε πέρα της δυσκολίας να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα. Σαΐντ κάνεις πολύ καλή δουλειά, το έχουμε συζητήσει. Θα είμαστε συνεργάσιμοι, θα υποβάλουμε τροπολογίες και θα είμαστε αποφασιστικοί, θα το κάνουμε μέχρι τέλους βάσει αυτού που είπε ο συντονιστής μου και η συγγήτριά μας, η σκιώδηση συγγήτρια. Όμως θα είμαστε σταθεροί και αποφασιστικοί όσον αφορά της, την αρχή μας ότι δεν θα πρέπει να τα φορτώνουμε όλα στην ε, συγκεκριμένη στην κατηγορία. Ο κύριος Φιντάντζα έχει το λόγο για ένα τρίλεπτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να τηρήσω το χρόνο μου, να παραμείνω στο χρόνο μου. Δεν έχω να προσθέσω πολλά περισσότερα σε αυτά που ήδη είπαν οι συνάδελφοι. Συμφωνώ με τη βασική αρχή που περιέγραψε ο κ. Δεγκράντες, δηλαδή τη θέση την ιδιαίτερη στην οποία βρίσκονται οι εκπρόσωποι των περιφερειακών χωρών όπου αντιμετωπίζεται μια δυσκολία στον αφορά την πρόσβαση στην κεντρική Ευρώπη, θα ήθελα να επισημάνω κάποια ε, σημεία δυσκολίες που παραμένουν. Αφήνοντας τις θετικές πτυχές επί των οποίων υπάρχει Γενική Συμφωνία. Το πρώτο θέμα λοιπόν είναι του mark-up και των διευρυμένων διαδρόμων. Πιστεύω ότι η αρχική εκδοχή ε, έδινε μια έναν ορισμό των διευρυμένων διαδρόμων πάρα πολύ ευρύ. Δεν ήταν στόχο η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά να ξεφορτωθεί το, να φορτώσουμε το κόστος στις περιφερειακές χώρες, αυξάνοντας την ανταγωνιστική δυσχερή του θέση. Και σαν δικαιολογία χρησιμοποιείται η μείωση του, των συνεπειών για το περιβάλλον. Είναι μια νέα διατύπωση. Εξετίμησα τα όσα είπε η συνάδελφος Βόρτμαν Κόλ, που ήθελε θέλει να εισάγει το θέμα της γειτονίας όσον αφορά τις παράλληλες διαδρομές, το καλύτερο θα ήταν να τα αφήσουμε όλα αυτά εκτός και να επιστρέψουμε στην αρχική, ε, στον αρχικό ορισμό. διάδρομος είναι διάδρομος και δεν υπάρχουν παράλληλοι δρόμοι και διάδρομοι. Όσον αφορά το θέμα των ε, διοδίων και το θέμα και πώς συνδέεται με το markup, νομίζω ότι αντιμετωπίζουμε μια θέση πολύ εύθραυστη σε σχέση με το Συμβούλιο. Και για να γίνει μια ανταλλαγή θα πρέπει να εξαιρεθεί το Euro 3 από τις κατηγορίες που υπόκεινται στο ποσό του markup με τα διόδια. Όσον αφορά τη διαμόρφωση του τέλους ε, της συμφόρησης δεν ξέρω αν πρέπει να αυξήσουμε τον πύχη το 150% του Συμβουλίου νομίζω ότι είναι κάτι που είναι πολύ επιβαρυντικό για τις επιχειρήσεις και μακριά από τις ανάγκες αγοράς. Δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε, πιστεύω, τον ορισμό, το σημείο συμβιβασμού του Συμβουλίου. Γιατί νομίζω ότι αυτή η θέση του Συμβουλίου είναι πολύ υψηλή. Και υπάρχει κάτι άλλο το οποίο δεν τα άκουσα να αναφέρεται από τους συναδέλφους αλλά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το ρόλο του Κοινοβουλίου. Είναι αυτό τον κατεξουσιοδότηση πράξεων. Το κείμενο που αναλύουμε θα έπρεπε να ενταχθεί, να επαναξαρθεί με όπως είναι το παράδειγμα 3 που αφορά τους υπολογισμούς. Θα μπορούσε αυτό να εξεταστεί με στον, τον κατεξοδότηση πράξεων. Θα πρέπει να υπάρχει, να ακολουθηθεί συνηθισμένη διαδικασία νομοθετική και τέτοια νομοθεσία δεν θα πρέπει να μπαίνει, να εντάσσεται στις κατεξοδότηση πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όσον αφορά το θέμα της αναθεώρησης της οδηγίας και την προσθήκη και άλλων εξωτερικών δαπανών που ήδη αναφέρονται στο κείμενο, εγώ θα ήμουν πολύ προσεκτικός, διότι ήδη προβλέπουμε τώρα ότι στην ε, ανάλυση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ετοιμάσει όσον αφορά την εφαρμογή της Ευρωβινιέτας θα προβλέπεται και πρώτες αναθεωρήσεις οδηγίας με νέο εξωτερικό κόστος που ήδη έχει εντοπιστεί, με νέες διαπάνες και νομίζω ότι με αυτό ξεπερνάμε ε, τα όρια. Ευχαριστώ. Κυρία Ράνα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να είμαι σύντομη. Κατερίνα θα ήθελα και εγώ να ε, γκομιάσω τον που ήξερε να θα αρχίσει τι θα τον περίμενα στη συζήτηση όπως σημερινή και όπου υπάρχουν τόσο τόσο διαφορετικές και αποκλίνουσες απόψεις. Τώρα που ξέρω έχω δει την, ε, την ε, οδηγία αυτή γραπτά, ίσως είμαι λιγότερο έτσι ενοχλημένη από τους ε, συναδέλφους, γιατί εγώ τη βλέπω πρώτη φορά και οι συνάδελφοι εργάζονται πολλά χρόνια πάνω στην Ευρωβινιέτα. δεν θα πρέπει να προσπαθήσουμε την σύγκρουση με το Συμβούλιο, από την άλλη μεριά ίσως να ξεκινήσουμε από μέγιστες απαιτήσεις για να συμφωνήσουμε πάνω σε έναν αποδεκτό συμβιβασμό. Μετά προστασία του περιβάλλοντος έχουμε βέβαια την ανάγκη της ε, ε, προσαρμογής των οικονομικών μας προβλημάτων με την προστασία των παραδείγματο χάρη ορεινών και Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο αυτή την εποχή να το πετύχουμε. Ελπίζω όμως ότι θα μπορέσουμε με αυτό που θα αποφύσουμε να μειωθεί η επιβάλληση του περιβάλλοντος με τα... από τα φερτηγά, ε, κάτι που αφορά και πάρα πολύ τη δική μου κυβέρνηση στην Αυστρία και θα ήθελα να τα κάτω κλιμάκια 0 έως 3 των φορτηγών θα πρέπει να ε, ληφθούν υπόψη ίσως με την ε, Ευρω 6 προχωρήσουμε κάπως περισσότερο και ίσως αυτό είναι κάτι που μπορούμε να επιβάλλουμε και στο Συμβούλιο. Αυτά είναι τα κύρια θέματα που μας αφορούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ρόνερ. Ο κύριος Κουμουτσάκος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Όσον αφορά το, το όνομά μου, είναι σίγουρα δυσκολότερο από το Σίμψον, αλλά πιστέψτε μου ότι για τους Έλληνες είναι το ίδιο πολύπλοκο με το Λίχτενμπέργκερ. Ευχαριστώ πολύ τον ε, εισηγητή για τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα, κύριε Πρόεδρε. Και θέλω να εκφράσω με αυτήν την ευκαιρία και τη συμπάθειά μου για το πολύ δύσκολο και πολύπλοκο έργο που είχε αναλάβει. Ε, επειδή έχουν τοποθετηθεί ε, συνάδελφοι. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος και θα μένω σε τρία μόνο σημεία. Πρώτον, ε, υποστηρίζω, θέλω να πω, την βασική φιλοσοφία των παρατηρήσεων του κ. Ντεγκράντες, ε, ειδικά για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν περιφερειακές χώρες με το μεγάλο συμπληρωματικό κόστος. Το δεύτερο σημείο είναι ότι είναι θετική η πρόνοια που υπάρχει για την επανεπένδυση στον τομέα των μεταφορών. Η τροπολογία 18 είναι μια θετική τροπολογία. Τέλος και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, για να μην παρατείνω μια συζήτηση που είναι ήδη μακρά. Θέλω να αναφερθώ ε, σε, σε μια συγκεκριμένη τροπολογία, στην τροπολογία 1 και ειδικά στο σημείο που αναφέρεται στις θαλάσσιες μεταφορές και την προβλεπόμενη από την τροπολογία συμπερίληψή του στο ETS. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να είμαι ξεκάθαρος εδώ. Πιστεύω ότι πρόκειται σαφώς για μία άσχετη με το χαρακτήρα και την στόχευση της οδηγίας αναφορά. Επιπλέον προκαλεί τουλάχιστον απορία για ποιο λόγο προβλέπεται ότι μια τέτοια συμπερίληψη θα γίνει και μάλιστα γρήγορα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, τίποτα άλλο. Thank you for the commission, Mr. Ευχαριστώ της Κομισιόν, κύριε Σμίτ. Σα schönen Dank. Äh, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πάρα πολύ καλή και επιμελή εργασία που επιτέλεσε για τόσο δύσκολη αυτή η πρόταση για την εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους. Θα ήθελα να ότι από πλευρά Κομισιόν και εμεί θεωρούμε ότι η ρεαλιστική προσέγγιση του κυρίου Αλκατράου είναι ακριβώ η σωστή. Πιστεύουμε ότι έχει φτάσει το πλήρωμα του χρόνου για να εφαρμόσουμε τι αρχέ στην πράξη και γλίγορα για να μπορέσουμε την θεωρία να την εφαρμόσουμε στην καθημερινή ζωή των οδικών μεταφορών. Γι' αυτό είναι αισιόδοξη η Κομισιόν ότι παρόλε τι αποκλίνουσε απόψει που ακούσαμε σήμερα, θα μπορέσει να επιτευχθεί καλό συμβιβασμό στη δεύτερη ανάγνωση. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, γι' αυτό θα περιοριστώ σε κάποια τεχνική μορφή ε, ερωτήματα. Ε, πέντε σημεία έχω σημειώσει. Καταρχήν η διαλειτουργικότητα. Είναι ένα θέμα που αναφέρθηκε πλειστάκι και θα ήθελα να ε, επιβεβαιώσω ότι και εμείς ε, στην Κομισιόν συμμεριζόμαστε τις επιφυλάξεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή όσον αφορά την λειτουργικότητα. Και βλέπουμε ότι είναι απαραίτητο και η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να ασχοληθούν εις βάθος με το θέμα αυτό, ούτω ώστε η εν λόγω οδηγία να μπορεί να οριστικοποιηθεί και να εφαρμοστεί. Συμφωνούμε λοιπόν απόλυτα με τροπολογία υπαριθμών 7 ίσως θα πρέπει να ε, βελτιώσουμε κάπως κάποιες διατυπώσεις, αλλά καταρχήν συμφωνούμε. Επίσης, η Κομισιόν θεωρεί ότι αυτό που προβλέπει το Κοινοβούλιο για να υπάρχει ουδετερότητα όσον αφορά τα, τα έσοδα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό θα βοηθήσει στην πράξη να... Ε, μπορέσουν οι μεταφορείς να έχουν τα σωστά μηνύματα και να μην ε, υπάρχουν έντονες διακοιμάσεις. Υποστηρίζει η Κομισιόν λοιπόν τις τροπολογίες 5 και 15. Όσον αφορά τώρα τη σύγκριση με άλλους ε, τομείς μεταφορών, Ξέρετε ότι για την Κομισιόν το θέμα αυτό του κόστους μεταφοράς δεν είναι μόνο θέμα της ε, αλήθειας όσον αφορά το κόστος αυτό του καθ' αλλά και μία μέθοδος για, την e, ευφυή, για τον ευφυή e προσανατολισμό των μεταφορών. Σε μερικέ εβδομάδε θα αρχίσει η συζήτηση για τη Λευκή Βίβλο και θα δείτε ότι πάνω σε αυτό θα ε, απαντηθούν πολλά από τα ερωτήματα που σήμερα παραμένουν ανοιχτά. Συμφωνούμε λοιπόν με πολλά από τα σχόλια που έγιναν και επίσης αυτά που αναφέρονται με την ε, στις τροπολογίες 23, 24, 26 που θα πρέπει να εξεταστούν υπό το φως της Λευκής Βίβλου κατά πόσον είναι ακόμα απαραίτητα. Επίσης, χαιρετίζουμε ότι το Κοινοβούλιο καλεί την Κομισιό να υποβάλει μια νομοθετική πράξη. Αναφέρομαι εδώ στην ε, τροπολογία υπαριθμών 25 σας παρακαλώ όμως να μην ξεχνάτε ότι πρέπει να σεβαστείτε το ε, δικαίωμα πρωτο, ε, πρωτοβουλίας της Κομισιόν και γι' αυτό να υπάρχει στα αγγλικά η διατύπωση if appropriate, εάν είναι κατάλληλο. Κατόπιν, θα αναφερθώ στην τροπολογία υπεριθμών 17 που λέγεται ότι ενδεχομένο πλεόνασμα εσόδων θα πρέπει να αντισταθμιστεί μέσα σε ένα έτος από πρώτης ματιάς δεν υπάρχει ένα τεχνικό διοικητικό πρόβλημα, αλλά ίσως υπάρχει ένα αρνητικό στοιχείο, δηλαδή διακοιμάνσεις της συγκυρίας θα α, μεταβάζονται άμεσα στον κλάθο και αν δείτε ας πούμε το έτος 2009 όπου γενικά ο αριθμός των οχημάτων που έπρεπε να πληρώνουν τα διόδια αυτά μειώθηκε σημαντικά, αυτό θα σήμαινε ότι εκείνο το έτος θα έπρεπε να αυξηθεί αμέσως το ύψος των διοδίων. Και γι' αυτό αυτή η μείωση από 2 στα 1, ε, τι όπως προβλέπετε στην τροπολογία και αυτά, φαίνεται ότι θα είναι πολύ υπαβαρυντική για τους ενδιαφερόμενους μου. Θεωρούμε ότι ο συμβασμός που επετεύχθη μετά από προσεπτικές εργασίες το 2006 είναι πολύ ευφυής ε, γιατί λέει ότι οι συνδυακές διακοιμάνσεις θα πρέπει να εξισωθούν και να μην οδηγούν αμέσως σε ψηλότερη επιβάρυνση του κλάδου. Λοιπόν, με αυτή την τροπολογία δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Και τεχνικά είναι τελικά συγγνώμη, ένα θέμα που δεν είναι τόσο τεχνικό ίσως, αλλά σημαντικό για την όλη συζήτηση. Δηλαδή, της δέσμευσης των πόρων αυτών για κάποιο συγκεκριμένο στόχο, της προσημείωσης δηλαδή των εξόδων. Ξέρει το σώμα ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Κομισιόν. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν εδώ δυσκολίες. Τι φάνηκε από τη συζήτηση και θεωρούμε ότι μια πραγματιστική προσέγγιση όπως αυτή που ακολουθεί ο εισηγητής είναι πάρα πολύ σοφή. Έχουμε το προηγούμενο με την οδηγία για το εμπόριο των εκπομπών όπου τονίζει ιδιαίτερα το θέμα της δημιουργίας διαφάνειας. Στην οδηγία αυτή για τις ε, εκπομπές ε, λέγεται ότι για τα έσοδα και για τις δαπάνες των, ε, από τις πωλήσει αυτές των εκπομπών θα πρέπει να υπάρχει μια απογραφή. Και μας φαίνεται ότι αυτό είναι πάρα πολύ καλό και αυτό θα πρέπει να βοηθήσει προτού αποφασίσουμε το θέμα της ε, προσημείωσης των εξόδων. Ελπίζω με τις παρατηρήσεις αυτές να απάντησα σε κάποια από τα ανοιχτά ερωτήματα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Σμίτ. Ο κύριος Αλκαντράουι, θέλετε κάτι να προσθέσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι Πολύ σύντομος. Ακούσαμε τους συναδέλφους και ένα ευρύ φάσμα απόψεων. Δεν είναι εύκολο να ικανοποιήσουμε τους πάντες, γιατί όταν θέλουμε να είμαστε πολύ φιλόδοξοι, ο καθένας διεκδικεί όλο και περισσότερα, αλλά δεν συμπίπτουν δυστυχώς οι διεκδικήσεις μας πάντα. Υπάρχει τέτοια διαφοροποίηση των απόψεων που είναι πολύ δύσκολη η επίτευξη σύγκληση ακόμη και στο Συμβούλιο. Ξέρατε τη θέση μου στην πρώτη ανάγνωση. Υπάρχουν κάποιες σαφείς απόψεις ό,τι αφορά την ε, εξωτερήκευση του κόστους, αλλά στην πρώτη ανάγνωση δεν συμφωνήσαμε με το Συμβούλιο προς αυτό. Με την εσωτερήκευση, συγγνώμη, του κόστους. Τώρα, για τα ποσοστά ή το συντελεστή των τελών. Να δούμε πώς μπορούμε να είμαστε ρεαλιστικοί. Η σημερινή πρόταση μιλά για κάποιο τέλος των υποδομών και εκεί θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή διαφοροποίηση, δηλαδή να δώσουμε στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να διαρθρώσουν καλύτερα και να διαχειριστούν την ροή των μεταφορών. Αλλά στα περισσότερα κράτη-μέλη σήμερα υπάρχουν τεράστια περιθώρια λιγμών σε ό,τι αφορά το τέλος των υποδομών και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να απολαμβάνουν αυτό το περιθώριο λιγμών. Σε ό,τι αφορά τον, την εσωτερήκευση του εξωτερικού κόστους, θα πρέπει να προβούμε στον κατάλληλο καταλογισμό ε, σε ό,τι αφορά την ε, ατμοσφαιρική ρήπανση, αλλά μην ξεχνάμε και την ηχορύπανση. Και αυτό το κόστος θα πρέπει κάπως να καταλογιστεί. το Συμβούλιο δεν μείωσε τα, τα ποσοστά σε ό,τι αφορά την ηχορύπανση. Αντίθετα τα αύξησε κάπως για να λάβει υπόψη την πραγματική κατάσταση. Και έχουμε και το θέμα του περιθωρίου σε ό,τι αφορά την προσάυξη που μπορεί να συνδυαστεί με την εισφορά των εισφορών και την εσωτερήκευση για τις πιο ρηπογόνες κατηγορίες οχημάτων. Και έχουμε και μια νέα προσέγγιση για τον για την επανεπένδυση που θα εξασφαλίσει μια μεγαλύτερη βιωσιμότητα των συστημάτων μεταφορών. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες, να διευκρινίσουμε, να συγκεκριμενοποιήσουμε ορισμένες διατυπώσεις. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας. Αλλά μην ξεχνάτε ότι εδώ θεσπίζουμε ένα πλαίσιο που δίνει διάφορες δυνατότητες και περιθώριο λοιμό στα κράτη-μέλη. Κάθε κράτος θα χρησιμοποιήσει διαφορετική γκάμα δυνατοτήτων. Εμάς μας ενδιαφέρει να προσδιορίσουμε αυτό το πλαίσιο το συντομότερο δυνατόν, ώστε να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν τα κράτη-μέλη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και μακροπρόθεσμα θα μπορέσουμε ίσως να διευρύνουμε αυτό το πλαίσιο και να καταλήξουμε ενδεχομένω και, και σε ένα ευρωπαϊκό σύστημα. Ευχαριστώ κύριε Αλκαντράη. Ο κ. Κουμουτσάκος έθεσε θέμα όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές een er Πρόκειται για την πρώτη τροπολογία. Εκεί αναφέρονται οι άλλοι τρόποι μεταφορά και για την εσωτερήκευση του κόστου ή άλλε προβλέψει που γίνονται. Οι ναυτιλιακέ μεταφορέ αναφέρονται αναφέρονται ως τομέας για τον οποίο θα μπορούσαμε να προβλέψουμε κάποιες αντίστοιχες διατάξεις. Εδώ θέλουμε να δώσουμε ένα γενικό πλαίσιο με όλες τις δυνατότητες, με ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων, γιατί αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα πλαίσιο για όλους τους τρόπους μεταφοράς, για όλα τα μέσα μεταφοράς και αυτό ζητήσαμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, Αν θέλετε να καταθέσετε τροπολογίες, ε, μην καθυστερήσετε, γιατί τον Απρίλιο θέλουμε στην Επιτροπή μας ε, να αποκρισταλώσουμε τη θέση μας και να την οριστικοποιήσουμε. Σίγουρα θα συνεχίσω τις επαφές με τους κοιόδης ηγητές και φυσικά θα συνεχιστούν και οι επαφές μας με το Συμβούλιο, ώστε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία που θα φέρνει το Συμβούλιο όσο πιο κοντά γίνεται στην συνενετική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν θα πρέπει να είμαστε υπερβολικά απαιτητικοί για να μην χρειαστεί μετά να κάνουμε και υπερβολικές υποχωρήσεις. Για να μην κάνουμε εμείς όλες τις υποχωρήσεις, αυτό είναι το σημαντικό. Ευχαριστώ. Σε πεθυμίσω ότι 18 Μαρτίου είναι η προθεσμία υποβολή ε, τροπολογιών ψηφοφορία στην Επιτροπή θα γίνει τον Απρίλιο και στην Ολομέλεια τον Ιούνιο. Προθεσμία για τροπολογίες 18 Μαρτίου. Ψηφοφορία στην Επιτροπή. Απρίλιο. Ψηφοφορία στην Ολομέλεια προβλέπεται τον Ιούνιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νέο σημείο τη ημερήσια διάταξη. Ολοκληρωμένη πολιτική όσον αφορά τι ε, μεταφορέ, Ο κ. Κουμουτσάκο είναι εισηγητή. Κύριε Κουμουτσάκο, πριν ξεκινήσετε, κύριε Κουμουτσάκο, να επενθυμίσω σ' όσου αναχωρούν, α αναχωρήσουν ήσυχα να επενθυμίσω και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι όλες οι συναντήσεις θα πρέπει να εξάγονται εκτός εθούσης και όχι εντός. Λοιπόν, σας παρακαλώ να μετακινηθείτε γρήγορα και ήσυχα.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 Κύριε Κουμουτσάκο. Η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική είναι μια νέα και δυναμική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασίζεται στην αντίληψη ότι μια αποτελεσματική πολιτική για τους ωκεανούς, τις θάλασσες, τις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές δεν μπορεί παρά να ακολουθεί μια συνολική, σφαιρική και επομένως διατομεακή προσέγγιση. Γι' αυτό και η κύρια επιδίωξη της ολοκληρωμένης θαλάσσια πολιτικής είναι να προωθήσει τον συντονισμό, την συνέργεια των επιμέρους πολιτικών που αφορούν στη θάλασσα. Στρατηγικός στόχος όλων αυτών είναι βέβαια το να μεγιστοποιηθεί το όφελος από μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη που θα είναι ευνοϊκή για όλους τους επιμέρους τομείς και τις πολιτικές με σεβασμό εννοείται στο περιβάλλον και με ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και συνοχής. Το κείμενο που συζητάμε σήμερα, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, είναι ο πρώτο χρηματοδοτικό κανονισμό για την υποστήριξη τη ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Ο πρώτο χρηματοδοτικό κανονισμό. Αφορά στην περίοδο 2011-2013 και το προβλεπόμενο ποσό είναι 50 εκατομμύρια ευρώ για αυτή την τριετία. Και σκοπό βεβαίω του κανονισμού είναι να συνεχιστεί και να εμπλουτιστεί και να, και να ε, ε, ενδυναμώσει τις προβαρασκευαστικές δράσεις και τα πιλωτικά σχέδια που υπήρξαν έως τώρα και υποστήριξαν την ανάπτυξη της ολοκληρωμένης θαλάσσης πολιτικής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μια σειρά από ψηφίσματα το 2007, το 2008 και το 2010 υποστήριξε και συνεχίζει να υποστηρίζει σταθερά την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Μάλιστα, στην πρόσφατη έκθεση, στο πρόσφατο ψήφισμα της κυρίας Μάισνερ, υποστήριξε και την χρηματοδότηση της πολιτικής αυτής με 50 εκατομμύρια ευρώ για το διάστημα 11-13. Όσον αφορά ορισμένα ειδικότερα ε, σημεία της πρότασης του κανονισμού που συζητάμε σήμερα, η νομική του βάση δεν μπορεί παρά να επηρεάζεται από τον οριζόντιο χαρακτήρα που έχει αυτή η πολιτική. Όσον αφορά το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ, πιστεύω ειλικρινά ότι είναι ένα μετριοπαθές, μικρό θα έλεγα ποσό, για τα δεδομένα της κοινοτική χρηματοδότησης πολιτικών. Εδώ θα μου επιτρέψετε μια επισήμανση. Η δυσχερής οικονομική συγκυρία και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί που πηγάζουν από αυτή δεν επιτρέπουν όμως την λογική των λευκών επιταγών ή μια άστοχη χρηματοδότηση δράσεων. Αυτό ήταν ένα από τα βασικά σημεία που μας απασχόλησε. Γι' αυτό και στο σχέδιο που παρουσιάζουμε φροντίσαμε πρώτον να εξειδικεύσουμε με τρόπο αναλυτικό αλλά και επαρκώς ευέλικτο τους γενικούς αλλά και τους ειδικότερου στόχους της χρηματοδότησης. Η τροπολογία, στην τροπολογία 8 περιγράφει ποιοι είναι αυτοί οι γενικοί στόχοι και τροπολογία που ακολουθεί τους επιχειρησιακούς όπως λέμε στόχους. Και αυτό για να είναι σαφές πού θα πάνε αυτά τα χρήματα. Ο δεύτερος, το δεύτερο στοιχείο ελέγχου της χρηματοδότησης ήταν το να αυξήσουμε το βαθμό του ελέγχου της εφαρμογής του κανονισμού με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι να ενισχύσουμε τις εκθέσεις πρόοδου και τις εκθέσεις αξιολόγησης της πορείας και της εφαρμογής του προγράμματος από την Επιτροπή. Είναι τροπολογία 26. Προβλέπετε μία έκθεση αξιολόγησης και ε, μία έκθεση πρόοδου και μία έκθεση αξιολόγησης. Ο δεύτερος τρόπος είναι να εισάγουμε την διαδικασία των πράξεων εξουσιοδότησης, της Delegated Acts, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης. Αναφέρομαι στις τροπολογίες 6 και 18. Κύριε Πρόεδρε, είναι μια διαδικασία που διασφαλίζει τον αποφασιστικό έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χωρίς να παραβλέπει την ανάγκη της απαραίτητης ευελιξίας κατά την εφαρμογή του προγράμματος. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι δίνεται ιδιαίτερη προτεραιότητα ώστε τα ωφέλη που θα προκύψουν από την ε, εφαρμογή να πηγαίνουν πρωτίστως στα κράτη-μέλη και στην Ένωση, χωρίς όμως να υποβαθμίζεται και η σκοπιμότητα της συνεργασίας με τρίτα κράτη. Εδώ θέλω να υπογραμμίσω κάτι. Η συνεργασία με τα τρίτα κράτη, ειδικά στα θέματα της θάλασσας, δεν μπορεί παρά να γίνουν στη βάση του σεβασμού του κοινοτικού κεκτημένου και στο πλαίσιο αυτό ειδικό βάρος έχει η στέρεη νόμιμη βάση για διεθνή συνεργασία που δίνει η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας και οι συναφές και οι συναφείς με αυτό διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις. Όσον αφορά την δημοσιο... τους δημοσιονομικούς πόρους που διατίθεται στο πρόγραμμα για τρέχουσα περίοδο, η πρότασή μας κάνει αναφορά στα όρια του κεφαλαίου 2, τα Margins Heading 2, που αφορά την διατήρηση και διαχείριση φυσικών πόρων. Καταλήξαμε σε αυτή την πρόταση γιατί είναι σύμφωνη και με τη λογική της γνωμοδότησης της Επιτροπής Προϋπολογισμού, Budget, Budget Committee, αλλά και της Επιτροπής Αλίας, η οποία έχει και εκείνη ε, προτείνει αυτή την κατεύθυνση. Κατά πόσον, το κατά πόσον η συγκεκριμένη πρόταση θα μείνει ως έχει, δηλαδή τα margins του heading 2 ως έχει, ή θα αλλάξει, θα εξαρτηθεί κατά πολύ από την πορεία των συζητήσεων από εδώ και πέρα. Επίσης πιστεύω ότι πρέπει και θα το προτείνω στη συνέχεια της διαδικασίας Πιστεύω ότι πρέπει να ενταχθεί η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στις δημοσιονομικές προοπτικές του 2013-2020. Με αυτή την αφορμή και επειδή μίλησα για την συμβολή άλλων επιτροπών θέλω να ευχαριστήσω ε, τις ε, άλλες επιτροπές, την Επιτροπή Περιβάλλοντος, την Επιτροπή της, ε, την Περιφερειακής Ανάπτυξης, την Επιτροπή του Προπολογισμού και βεβαίως ιδιαίτερα την Επιτροπή Αλίας για την συνεργασία που είχαμε, για την ε, ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων και για τις γνωμοδοτήσεις τους βέβαια, στοιχεία από τις οποίες έχω συμπεριλάβει στο ε, σχέδιο που σήμερα κατατίθεται και είναι μια διαδικασία που θα τη συνεχίσουμε και μετά. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους άντρους ραπορτές, ε, με τους οποίους θα συνεχίσουμε και στο επόμενο στάδιο της στενής συνεργασίας μας, με ανοιχτό μυαλό και επικοδομητική πιστεύω διάθεση. Τέλο, ιδιαίτερη μνήμα θέλω να κάνω στην Επιτροπή και στην κυρία ε, Μπενίνη για την συνεργασία που είχαμε, αλλά και σε συναδέλφου από το Συμβούλιο, με του οποίου είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψει, να μοιραστούμε προβληματισμού και ιδέε. Κλείνω με δύο σημαντικέ, πιστεύω, επισημάνσει. Το πρώτο έτος χρηματοδότηση του προγράμματος ήδη τρέχει. Είμαστε στο 2011. Ο χρόνος λοιπόν που έχουμε για να καταλήξουμε στον, ε, στον, ε, στον κανονισμό είναι περιορισμένος. Είναι εξαιρετικά περιορισμένος. Πρόθεσή μου είναι, και θα το επιδιώξω, να υπάρξει συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση. Και επίσης να λάβω υπόψη μου όσο το δυνατόν περισσότερο από τις τροπολογίες τα σχόλια των σκιωδών εισηγητών αλλά και των άλλων συναδέλφων. Με μία επισήμανση. Χωρίς όμω να μετατρέψω το συγκεκριμένο τεχνικό και το τεχνικό αυτό κείμενο, αυτόν τον χρηματοδοτικό κανονισμό, χωρίς να το μετατρέψω σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο με κάθε είδου στολίδια που όμως θα έχουν λίγη ή καθόλου σχέση με το χαρακτήρα, το περιεχόμενο και το στόχο του κανονισμού. Πιστεύω ότι μια ισχυρή θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ενισχύσει και τη δική μου διαπραγματευτική θέση στην, ε, στις συνομιλίες με το Συμβούλιο και κυρίως θέλω τη στήριξη των συναδέλφων όσον αφορά το ύψο του ποσού των 50 εκατομμυρίων ευρώ αλλά και τις delegated acts, γιατί θα αποδειχθούν στην πορεία, πιστεύω, τα δύο πιο ακαθόδη προβλήματα που πρέπει να λύσουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Thank you, Mr. Σας ευχαριστώ κύριε Κουμουτσάκο. Ευχαριστήσατε το Συμβούλιο, αλλά σαν Έλληνας δεν σας πειράζει να σας υπενθυμίσω το θέμα του δουρίου ύπου. Ήθελα να το αναφέρω το θέμα του δουρίου ύπου. Για το S&D ο κύριος Μιλάνα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κάναμε καλή δουλειά. Θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντας τον συνάδελφο εισηγητή με τον οποίο συναντηθήκα μερικές φορές και συμφωνήσαμε σε όλα τις θέσεις μας. Συζητούμε λοιπόν την ολοκληρωμένη α, θαλάσσια πολιτική και αυτό είναι το πλαίσιο. Συζητούμε πώς η εμπειρία των τελευταίων τριών ετών με μικρές χρηματοδοτήσεις θα εφαρμοστεί με τα 50 εκατομμύρια ευρώ που είναι υπόθεση. Είναι μεγάλο θέμα. Πολύ σημαντική συζήτηση. Δεν συζητάμε κάτι επαναστατικό. Θα χρειαζόταν πολλές, πολλοί άλλοι πόροι για να εφαρμόσουμε πραγματικά μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Ήταν κοινή προσπάθεια, κοινή δουλειά. μου ουσιαστικά όλες τις τοποθετήσεις που ακούστηκαν. Υπάρχουν ένα-δύο ζητήματα που κατά την άποψή μου θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικότερα. Είναι ανοιχτή συζήτηση. Ήταν ανοιχτή συζήτηση, το λέω με κάθε με ηρεμία όσον αφορά τις λεπτομέρειες επί των οποίων βασίζεται αυτό το κείμενο. Και εγώ και κάποιοι άλλοι έχουμε κάποιο πρόβλημα όσον αφορά την κατανομή των πόρων που είναι μόνο στο παράρτημα ε, αυτό δημιουργεί θα δημιουργήσω κάποια προβλήματα μετά στην εφαρμογή όσον αφορά τη θέση του Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή Προπολογισμών ήδη ενέκρινε κάποια σχετική τροπολογία. Γίνεται και συζήτηση στην Επιτροπή Αλία. Προβλέπεται εκεί ότι στον κανονισμό θα, θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη αυστηρότητα όσον αφορά τον προορισμό των πόρων και την κατανομή που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να αποφύγουμε μετά από αυτή τη συζήτηση να γίνει αποδυνάμωση ε, των στόχων των δαπανών και των πόρων. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχιστεί αυτός ο προβληματισμός Μέχρι σήμερα το πρωί υπήρχαν επίσημε επαφές με, με του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προτείνουν τεχνικές διευθετήσει διαφορετικές, Ούτω όσο ο στόχος του Κοινοβουλίου τελικά να γίνεται σεβαστό στο τέλος της διαδικασίας. Χρειάζεται να εξετάσουμε περισσότερο το θέμα που αυτή την τροπολογία που μεταφέρει από το παράρτημα στο διατακτικό του κειμένου και ίσω χρειάζεται καλύτερο ορισμό στα άρθρα 2 και 3 που καθορίζονται περισσότερο οι στόχοι των προγραμμάτων. Πέρα από αυτό, εκτό αυτού, αυτών των σκέψεων, το υπόλοιπο του κειμένου με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο και έχουμε το χρονοδιάγραμμα. Ο χρονοδιάγραμμα που σα στην Επιτροπή Αλίας δείχνει ότι ο χρόνο είναι πολύ περιορισμένο, πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα. σω μαζί με τον συγητή ε, μπορούμε να το σκεφτούμε αυτό το θέμα και να δούμε πού μπορούμε να βοηθήσει. Ίσως η ιδέα των περιοδικών προγραμμάτων, των πιο επικέρων, ίσως να είναι μία λύση. Ένα άλλο στοιχείο, μία παρατήρηση για τροπολογία 11, που πρότεινε ο εισηγητής. Εγώ θα συμμεριζόμουν τον κατάλογο αυτών των θαλασσών. Υπάρχει πάντα περιθώριο όμως να λησμονηθεί κάποιο. Και αν υπάρχει κατάλογος με αναφορά θαλασσών και περιοχών, ο κίνδυνος είναι ίσως αυτός ο κατάλογος ε, να έχει αφήσει εκτός κάτι. Στην τροπολογία 10 δεν κατάλαβα καλά γιατί ε, ξερέτε με τους διάφορους ε, διαφερούμενους φορείς η συζήτηση και επαφή. Τελευταία παρατήρηση είναι το θέμα της Μεσογείου η Μεσόγειος είναι ο τόπος προνομιούχος για την εφαρμογή εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως πολιτικών ολοκληρωμένων για τις θάλασσες. Διότι ε, υπάρχουν 7 ευρωπαϊκές χώρες και καμιά δεκαριά και ανήσυχε μάλλον που υπάρχουν ταραχές χώρες εκτός Ευρωπαϊκής. Αυτό δείχνουν αυτά που συμβαίνουν τώρα. Υπάρχουν προβλήματα ρήπανσης αυτή τη θάλασσα στη Μεσόγειο, προβλήματα μεταφορών πολύ συχνά. Υπενθυμίζω ότι είναι η περιοχή με τη μεγαλύτερη παράκτεια δραστηριότητα όλης της, σε όλη την Ευρώπη. Αυτή η θάλασσα πραγματικά εκεί χρειάζεται αυτήν την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και χρειάζονται επαφές πολύ περισσότερες ε, με τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Όπω και στον Εύξηνο Πόντο έχουμε τρει χώρε Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής τέσσερι τέσσερις μη. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση για τον καθορισμό πιλωτικών προγραμμάτων ή καλύτερο ορισμό, ορισμού στα άρθρα 2 και 3, να εμπλουτίσουμε το κείμενο και να βρούμε σωστή προσέγγιση κατά τα λοιπά. Πιστεύω ότι είναι περιορισμένο το χρονοδιάγραμμα, είναι κάπως ορισμένη χρόνη. Πριν μου αφαιρέσει λοιπόν το λόγο ο Πρόεδρος, σταματάω. Σας ευχαριστώ κυρία Μάισνερ για Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν πρόκειται για ένα θέμα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ, το ξέρουν όλοι και γι' αυτό λυπούμε που δεν είναι γεμάτη η Γιατί φύγανε τόσο πολύ μετά την Ευρωβινιέτα. Ίσως επειδή δεν διακυβεύονται τόσο πολλά χρήματα και δεν είναι τόσο γνωστή η ολοκληρωμένη θανάσια πολιτική. Όλα αυτά μπορούν να βελτιωθούν βέβαια. Αυτή είναι μια εισαγωγική παρατήρηση. Δεύτερη εισαγωγική παρατήρηση. Και εγώ θα πρέπει να φύγω σε λίγο. Γιατί αυτή τη στιγμή εργάζομαι εκ παραλλήλου σε δύο επιτροπέ. Θα μου πούνε βέβαια αυτό που ελέγχθη. Συμβαίνει αυτό. Τώρα, όσον αφορά αυτή καθ' την έκθεση. Είπα ήδη. Από δική μου σκοπιά είναι μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση. Πρόκειται για μόνο 50 εκατομμύρια ευρώ, αλλά για 50 εκατομμύρια ευρώ που θα πρέπει λογικά να χρησιμοποιηθούμε προς όφελος των κρατών μελών και προς όφελος της Ευρωπαϊκής πολιτικές Πολιτικής. Και υπήρχε και κάποια φήμη ότι αυτά τα 50 εκατομμύρια διακυβεύονται, ότι θα μειωθούν. Γι' αυτό προσπάθησα να το ε, βρω αυτό αν ήταν αληθές, γιατί υπήρχαν τρεις προτάσεις. Να μην δοθεί τίποτα, να δοθεί κάτι, 50 εκατομμύρια ή πάρα πολλά χρήματα που δεν ήταν δυνατόν, αλλά ευκταίο. Θα πρέπει τα χρήματα αυτά να δαπανηθούν όσο δυνατόν πιο αποτελεσματικά γίνεται. Ξέρω ότι η Επιτροπή Προπολισμών έχει, υποβάλει, έχει προετοιμάσει ήδη μια γνωμοδότηση, σήμερα νομίζω ψηφίζουν επ' αυτής, όπου υπήρχε κάποια θέση 33 εκατομμύρια γενικά για ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική χωρίς λεπτομέρειες. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες ανοιχτές. Ταυτόχρονα η Κομισιόν έχει υποβάλει πάρα πολλές προτάσεις. Λοιπόν, ε, θεωρώ ότι η έκθεση είναι πάρα πολύ καλή. Ιδίω ε, θεωρώ πολύ καλό ότι ο κ. Κουμουτσάκος με τον οποίο συνεργάστηκα και πάνω στη δική μου έκθεση, ότι ο κ. Κουμουτσάκος λέει μπαίνει λεπτομέρειες και στην λειτουργικότητα της πρότασης ε, προσπάθησε να αναφερθεί συγκεκριμένα σε δράσεις. Είναι πιο ενεργή δηλαδή πια η έκθεση και μου φαίνεται πάρα πολύ καλό. Αναφέρθηκε επίσης πώς θα πρέπει ακριβώς να προχωρήσουμε και γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ευθυγραμμισμένοι. Λίγα πράγματα είναι αυτά που θα ήθελα να παρατηρήσω πάνω στις ε, τροπολογίες του κυρίου Κομουτσάκου. Καταρχήν τροπολογία υπ. 4, δεν ξέρω ίσως οφείλεται ο, στην μετάφραση του κοινού μου, είναι οι ομάδα των ενδιαφερομένων διαγράφονται. Δεν ξέρω γιατί. Εγώ νομίζω ότι πρέπει πάντα να αναφέρονται. Ίσως καμιά φορά χάθηκε αυτό στην μετάφραση του κειμένου. Το ίδιο και για την τροπολογία υπεριθμών 8, όπου δεν αναφέρονται πια οι παράκτιες περιοχές. Καλό είναι να αναφέρονται, παρόλο που εννοούνται ίσως. Και επίσης στην τροπολογία υπεριθμών 28 υπάρχει μια σημαντικότητα καινοτομία. Καταρχήν, λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συνοδευτική επιτροπή, αλλά με κατεξοικειοδότηση πράξης. Αλλά υπάρχει το θέμα της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων. Δεν ξέρω, μήπως εδώ έχουμε ένα ε, γκολ βάζουμε σε αυτούς μας κατά κάποιον τρόπο αυτό θα πρέπει ίσως να το εξετάσουμε καλύτερα, να το συζητήσουμε πώς θα λειτουργήσει το θέμα στην πράξη. Κατά τα άλλα μου φαίνονται πάρα πολύ καλά ότι ο εισηγητής σε όλα τα σημεία προσπάθησε να ε, δώσει μια πρακτική μορφή για τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου. Τέλος, όσον αφορά την Μεσόγειο, και ο κ. το είπε αυτό, είναι πολύ ενδεδειγμένη η Μεσόγειος για να υπάρχει μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική γιατί είναι πολύ μεγάλη θάλασσα, ε, είναι γύρω τόσα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, υπάρχουν προβλήματα μόλις, το είπε και ο αυτό, αλλά βέβαια θα πρέπει οι πόροι που έχουμε να καταναμηθούν στην Ευρώπη. Γιατί θα μπορούσαμε ίσως ε, για τη Μεσόγειο και μόνο σε πολλά σχέδια να δαπανίσουμε εκάστοτε 50 εκατομμύρια και αυτό δεν επιτρέπεται βέβαια γιατί τελικά για να μπορεί να είναι αποδεκτό το σύστημα αυτό, η πρόταση αυτή που προτείνεται, όλοι θα πρέπει να έχουν εντύπωση ότι ωφελήθηκε η χώρα τους. Αυτά και θα χαρώ για τις περαιτέρω συνόμες διαπραγματεύσεις της έκθεσης. Σας ευχαριστώ βέβαια, δεν το είπα ακόμα, στον συνάδελφο Κουμουτσάκο για την έκθεσή του. Ευχαριστώ και δυστυχώς πρέπει να φύγω τώρα. Hey, thank Σας ευχαριστούμε, ο κύριος ε, Τέιλερ από τους Πράσινους. Ευχαριστώ. Και εγώ δυστυχώς αμέσως μετά την παρέμβασή μου θα χρειαστεί να φύγω. Πάντως ήθελα καταρχήν να καθησυχάσω τον κύριο Κουμουτσάκο ότι οι πράσινοι θα υποστηρίξουν τα 50 εκατομμύρια ευρώ για την επόμενη διετία. Η τροπολογία δείχνει ότι τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για πολιτική, διακυβέρνηση, βιωσιμότητα και εποπτεία και νομίζω ότι αυτό ως πρώτο βήμα είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο. Εξετάζοντας ε, συνολικά την έκθεση, διαπιστώνω ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου χαιρετίζει ορισμένες από τις εξελίξεις που ε, θεωρούν ότι επιφέρουν προστιθέμενη αξία. Βέβαια δεν θέλουν να βάλω το χέρι στην τσέπη η Βρετανία, αλλά την προστιθέμενη αξία την καλωσορίζουν. Επίσης η προστιθέμενη αξία έγκυται σε διάφορα χειρά μηνύματα διασταυρωμένα και πολυεπίπεδα και νομίζω ότι θα πρέπει να ξανασκεφτούμε και το θέμα των περιβαλλοντικών κλιματικών αλλαγών και της ενεργειακής πολιτικής. Γιατί η ομάδα μου την οποία εκπροσωπώ εδώ και ο για το θέμα αυτό, θεωρεί ότι έχουμε την ευκαιρία να καθορίσουμε πραγματικά φιλόδοξους στόχους και στο θέμα της πολιτικής για τις κλιματικές αλλαγές. Στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε για την Ευρωβινιέτα, ακούσαμε την Επιτροπή να αναγνωρίζει την ανάγκη για μείωση των εκπομπών του διοξίδιου του άνθρακα σε όλες α, τους τρόπους μεταφοράς. Και με τις τροπολογίες που θα καταθέσουμε, θα προσθέσουμε τη συμπερίληψη των θαλάσσιων μεταφορών στο σύστημα εμπορίας εκπομπών. Πάντως και για τα θέματα κλιματικών αλλαγών και γενικότερη ρήπανσης θέλουμε τροπολογίες για καθαρότερους κινητήρες, καθαρότερα καύσιμα, καθαρότερα πλοία και επίσης ε, κάποιες απόπειρες για την αντιμετώπιση του προβλήματος του μαύρου άνθρακα αναφέρονται και ισχύουσες οδηγίες για το, τον έλεγχο του κράτους λιμένα, για τον έλεγχο των, της κυκλοφορίας και τη διαλεύκανση μάτων. Βέβαια, το θέμα αυτό το καλύψαμε εν μέρη και στην πρόσφατη έκθεση της κυρίας Μάισνερ, το θέμα των, της παραγωγής πετρελαίου offshore, γιατί είδαμε ότι πολλές φορές ε, η φύση μπορεί να έχει τρεις συνέπειες. Είδατε τι έγινε με την Ιαπωνία και είδαμε και το ατύχημα στον κόλπο του Μεξικού. Νομίζω ότι από τα παθήματα αυτά θα πρέπει να αντλήσουμε κάποια διδάγματα και επίσης να δούμε και το θέμα της μεταφοράς επικίνδυνων υλικών, ιδιαίτερα από ευαίσθητες θαλάσσιες περιοχές και υπάρχει και το θέμα επίσης του καμποτάζ των παράκτιων μεταφορών. Ίσως καλό θα ήταν ε, χρησιμοποιώντας καλύτερες αλλάσεις μεταφορές να ελαφρύνουμε κάπως τις οδικές μεταφορές. Θα συμβάλλουμε στην ε, ανάπτυξη αυτής της συνέκθεσης και ευχαριστούμε και πάλι τον εισηγητή για τη μέχρι τώρα προεργασία που έκανε. Ο κύριος Βαντάλεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή μας, ο οποίος ε, εκπώνησε μια αξιόλογη έκθεση. Θα ήθελα να σταθώ λίγο στην τροπολογία 17, όπου ο εισηγητής διευκρινίζει ότι το πρόγραμμα αυτό θα παρέχεται μόνο εφόσον διατίθεται άλλη χρηματοδότηση από την Ένωση, σχετική χρηματοδοτική στήριξη. Σε τι αφορά τα σχόλια του κυρίου Μιλάνα για τη Μεσόγειο, αυτό που μας ενόχλησε ήταν ότι είπε ότι προσοχή να μην είμαστε υπερβολικά τολμηροί, υπερβολικά φιλόδοξοι, να μην προκαθορίζουμε ακόμη τη χρήση των κονδυλίων. Για παράδειγμα, σε ορισμένε τροπολογίε ο εισηγητή μα δίνει πολύ συγκεκριμένε προτάσει που δείχνει τι θέλουμε συγκεκριμένα. Εγώ θα προτιμούσα πιο γενικές εξαγγελίες ανάλογες με αυτές του κανονισμού. Εκεί θα, προσπαθήσουμε, θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια συμβαστική λύση. Σίγουρα οι τροπολογίες περιλαμβάνουν πολύ εύστοχα θέματα. Εμείς είχαμε παλιά μιλήσει για, τα, για τους πράσινους λιμένες και το θέμα της αηφορίας της ε, βιωσιμότητας και στους λιμένες. Το είχαμε θέσει παλιά ομάδα. Ε, καλό θα ήταν να επαναφέρουμε αυτή την ιδέα εδώ για να καταπολεμήσουμε τη μόλυνση, τη ρήπανση στους λιμένες. Θα καταθέσουμε λοιπόν μια τροπολογία με αυτή την ιδέα των πράσινων λιμένων. Εν κατακλείδη, θα ήθελα να υπενθυμίσω αυτό που είπατε για το δούριο ύπο σε σχέση με το Συμβούλιο. μην ξεχνάμε τι έγινε με, το, με τον Εννέα ε, και την ίδρυση της Ρώμης. Ε, μερικές φορές και από τέτοιες περιπτώσεις έχουμε πολύ αίσια αποτελέσματα. Ευχαριστώ κύριε Βαντάλεν. Εσείς και εγώ θα πρέπει να διαβάσουμε περισσότερο τον Τροϊκό Πόλεμο και την κυριαρχία των Αθηνών κλπ. Ο κύριος Ρίκια έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να συγχαρώ τον Γιώργο για τη δουλειά που έκανε. Σαν ε, εισηγητής για την Επιτροπή Προπολογισμών για τη στέξη γνωμοδότηση, θα ήθελα να κάνω κάποιες διευκρινήσεις και να σε κάποια σχόλια. Θα γίνει αύριο το πρωί ψηφοφορία στην Επιτροπή Προπολογισμών. Δεν έχουν ψηφίσει ακόμα. Στην Επιτροπή Προπολογισμών θέλαμε να περιοριστούμε στις πτυχές του προπολογισμού. Χωρίς να συζητήσουμε τις ουσίες, όπως ξέρεις Γιώργο. Λοιπόν, το πρώτο θέμα είναι τα 50 εκατομμύρια ευρώ, πώς θα μοιραστούν, το ποσό που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω που θα γίνει αποδεκτό το ποσό από την Επιτροπή Προπολογισμών εξασφαλίζοντας καλύτερη πλαισίωση και καλύτερο έλεγχο των δαπανών. Θα είμαι σύντομος. Στην Επιτροπή Προεπολογισμών υπογραμμίστηκε εν πρώτης πως ότι δεν θα πρέπει να γίνει χρηματοδότηση αυτής της πολιτικής εις βάρος άλλων πολιτικών. Έχουμε υποβάλει σχετική τροπολογία. Αυτά τα 50 εκατομμύρια ευρώ μπορούν να βγουν από το κεφάλαιο 2 από το αποθεματικό. Είναι σημαντικό θέμα, διότι ανησυχεί πολλούς. Μετά, θα πρέπει στην θέτηση του προγράμματος εργασίας να συμμετέχει το Κοινοβούλιο όσον αφορά το, τη χρηματοδότηση, τη χρηματοδότηση και τα ποσοστά θα πρέπει αυτά που αναφέρονται στο παράρτημα να μπουν στο διατακτικό. Αυτό δεν είναι ανέφικτο για λόγους τυπικούς. Το έκανα στην έκθεσή μου και αφού το συζήτησα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έγινε ο νομικός έλεγχος, θα το αφαιρέσουμε από το κείμενο. Δεν μπορεί αυτό το παράρτημα των δαπανών να μπει στο κυρίω κείμενο. Και γι' αυτό έβαλε αυτή την αναφορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο παράρτημα. Είναι ανέφικτο. Εξίσου, προτείναμε κονδύλια, γραμμές του προπολογισμού και αυτό είναι ανέφικτο διότι δημιουργούνται κατά την ψηφοφορία του προπολογισμού αυτές οι γραμμέ και υπό αυτέ τι συνθήκες δεν μπορούμε να αναφέρουμε σε πρώτερη έκθεση. Είτε είναι η έκθεση τη ουσία ή είτε η έκθεση της ε, επιτροπή Προπολογισμών. Είχε εκφραστεί με ανησυχία αυτό το λέω. Ότι ο καθορισμός των κονδυλίων δεν επηρεάζει καθόλου την αρμοδιότητα τη Επιτροπής. Αν τα κονδύλια ενταχθούν στην πολιτική αλίας αυτό δεν είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Μεταφορών επί της ουσίας. Σας το λέω. Δεν ήταν επί της συζήτηση όσον αφορά την, ε, τα κονδύλια του προπολογισμού, τις γραμμές του προπολογισμού. Η ενδιάμεση εξολόγηση της πολιτικής που πραγματοποιείται από το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό αναφέρεται το Γιώργο, και υπάρχει ένα πρόβλημα, είναι η βιωσιμότητα της χρηματοδότησης, θα γίνει μετά το 2013. Ψηφίζει αύριο η Επιτροπή, υπάρχει ευρεία συμφωνία για την έκθεση που υπευλήθη και θα συμπεριληφθεί με τις τροπολογίες στην βασική έκθεση του Γιώργου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Φώστερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Εν γέννη, υποστηρίζω τους βασικούς στόχους της εκθέσεως. Υπάρχουν ένα-δύο ερωτηματικά που έχω, που θα θέσω πιθανότατα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χρειάζεται κάποια προσοχή Όσον αφορά την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, θα πρέπει το πρόγραμμα να δείχνει ότι επιτυχάνει επωφελή αποτελέσματα, κυρίως το δύσκολο οικονομικό κλίμα. Αναφέρομαι και στις λογικές σκέψεις για τη χρηματοδότηση της σας. τα 50 εκατομμύρια που προτάθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύω ότι θα πρέπει να βγουν από υφιστάμενα κονδύλια Ίσως θα μπορούσε να το διευκρινίσει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από πού θα βγουν αυτά τα 50 εκατομμύρια, πού προέρχονται. Θα χρησιμοποιηθούν λοιπόν τα χρήματα, χρησιμοποιούνται τα χρήματα για προγράμματα και έργα και πρέπει να συζητηθεί η χρήση των πόρων. Και πώς θα γίνεται ο έλεγχος της χρήσης των κονδυλίων. Τα ανέφεραν και άλλοι συνάδελφοι της Επιτροπής. Για τις τροπολογίες 4 και 8 αιτιολογική σκέψη 6 και άρθρο 2 αφορούν. Θέλω διευκρίνηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την χρήση της λέξης εκτέλεση, υλοποίηση. Προβλέπεται μια ρυθμιστική διαδικασία που ίσως αντιβαίνει την επικουρικότητα. Μπορεί να το ξεκαθαρίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τροπολογία 12 που αφορά το άρθρο 3. Έχω πρόβλημα με τη χρήση της λέξης διασυνοριακή και αυτό σε σχέση με τις διασυνοριακές εποπτικές δραστηριότητες και διευκόλυνση διασυνοριακό, διασυνοριακής ε, θαλάσσιας χωροταξίας. Η χρήση της, του όρου διασυνοριακός ίσως να υπονομεύει την αρχή της επικουρικότητας. Εμπεριέχει πολλά καλά στοιχεία η έκθεση. Όπως σας είπα όμως, ο εισηγητής είπε ότι πρέπει να προχωρήσουμε και να πετύχουμε αποτελέσματα στην πρώτη ανάγνωση. Να θυμηθούμε όμως πρέπει ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τι υποχρεώσεις υπέχουμε σύμφωνα διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις και τα κρατημέλη. Άρα πρέπει να κινηθούμε σωστά. Ευχαριστώ εκ νέου τον εισηγητή και προσβλέπω στα σχόλια και τις διευκρινήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Κούν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και δεν ήθελα να ευχαριστώ και εγώ τον Γιώργο Κουμου, Κουμουτσακό, σωστά το είπα. Η περιγραφή ήταν πολύ καλή προηγουμένως. Υπάρχουν περισσότερα μέλη εδώ από χώρες που δεν έχουν καθόλου πρόσβαση στη θάλασσα όπως η και ο συνάδελφος εδώ και που ενδιαφέρεται όμως να υπάρχει μια κοινή ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Γιατί βέβαια αυτό αφορά την κοινή μας εσωτερική αγορά. Και όλοι οι ύφαλοι για του οποίου έχουμε συστήσει εδώ πολλές φορέ στην Επιτροπή Μεταφορών παίζουν σημαντικό ρόλο. Τα διευρωπαϊκά δίκτυα, παραδείγματο χάνει, παίζουν σημαντικό ρόλο. Κατά μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό η στρατηγική αυτή να βασιστεί σε αυτά που γίνονται σήμερα περιφερειακά στις επιμέρους μακροπεριφέρειες που ανέφερε ο κ. Μιλάν. Να συνδεθούν αυτές οι διάφορες δραστηριότητες μεταξύ τους. Στρατηγική για τη Βαλτική έχουμε. Έχουμε στρατηγική για τον Ατλαντικό και για τη Βορειοθάλασσα. Έχουμε τη Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα. Όλα αυτά είναι δραστηριότητες που μπορούν να ενταχθούν μέσα στην γενική ε, επικεφαλίδα, αν θέλετε, ε, ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Έχουμε δηλαδή ένα θέμα χώρο ταξίας των θαλασσών. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό που ορίζεται στην πολιτική και ρωτώ την Κομισιόν τώρα Όταν με αυτό το πενιχρό ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ προσπαθούμε να εφαρμόσουμε την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, στα κράτη-μέλη, ποια είναι η δική σας εμπειρία, αν από, τα, από τη Μεσόγειο, πούμε, τα διάφορα κράτη-μέλη έχουν ομάδες εργασίας οι οποίες προσπαθούν αυτή τη χωροταξία να την προωθήσουν σε πλαίσια της οδηγίας πλαίσιο της στρατηγικής μας. Θα πρέπει να εξεταστούμε να εξετάσουμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε τους πόρους που έχουμε εδώ, τους θαλάσσιους. Θαλάσσιες μεταφορές, σπορτ, ε, σπορ, αθλητισμός, ε, ε, αλληλεία φυσικά πάρα πολύ σημαντικό, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η διαφραγωγή που χρειάζεται γι' αυτό μέσα στη θάλασσα κλπ. Και άμα συζητάμε για την κοινή ιστορική πολιτική θα πρέπει να έχουμε τα ίδια πρότυπα. τους όσον αφορά τι εκπομπέ καυσαερίων από τα πλοία ή και από τα λεγόμενα green parts. Και πώ θα συμπεριληφθούν χώρε που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω η Ρωσία ή οι χώρε τη Αυτά τα πρακτικά θέματα θα ήθελα να μου τα εξηγήσει η Κομισιόν, παρακαλώ ευχαριστώ. Ο κύριος Δανέλης, Πρόεδρε. Ε, βεβαίως περνάμε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, αλλά το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ για δύο χρόνια είναι ελάχιστο για τους σκοπούς που το θέλουμε και μικρό σχετικά για μια ευρωπαϊκή πολιτική. Ε, φαντάζομαι δε ότι ε, εφόσον όλοι εκτιμούμε ότι αυτή η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική πρέπει όλο και να ενισχύεται, δεν έχουμε άλλο τρόπο παρά να εντάξουμε την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στις δημοσιονομικές προοπτικές 13-20. Ε, μου αρέσει η ενίσχυση των ελέγχων χρηματοδότησης με συνεχείς εκθέσεις ελέγχου και αξιολόγησης, διότι αφενός εγγυάται την ορθολογική αξιοποίηση των ελάχιστων πόρων που διαθέτουμε, αφετέρου αναδεικνύει και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχει ένα ζήτημα εξασφάλισης ευελιξίας, ε, έτσι δεν ξέρω αν ε, οι πράξεις ε, εξουσιοδότησης είναι το κατάλληλο εργαλείο υπό αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να το εξετάσουμε παρότι όντως φαίνεται σαν δούριος ύπος. Νομίζω ότι θα πρέπει να θεωρούμε αυτονόητο ότι οι σχέσεις της Ένωσης με τις τρίτες χώρες, με τα τρίτα κράτη, θα πρέπει να βασίζονται στο κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα βέβαια στη συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας που αποτελεί και τη βάση του κράτους δικαίου για τις θάλασσες. Τέλος, ε, συμφωνώ ότι επειδή είναι ανάγκη να προχωρήσουμε και ουσιαστικά και γρήγορα έχουμε χάσει ήδη το μισό του πρώτου από τα δύο χρόνια, ε, θα πρέπει να περιοριστούμε στη συζήτησή μας ε, σε ό,τι αφορά την ουσία του χρηματοδοτικού αυτού κανονισμού και όχι οποιασδήποτε εκκρεμότητα έχουμε να ρυθμίσουμε σε σχέση με την θαλάσσια πολιτική συνολικότερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές για τη δουλειά που έκαναν. Θα ήθελα να πω ότι είναι ένα σημαντικό βήμα πάνω σε ένα θέμα που ήδη τους τελευταίους μήνες εξετάσαμε και το θέμα το αντιμετωπίζουμε τώρα δείχνει ότι συμμεριζόμαστε κατά πόσο είναι σημαντική αυτή η πολιτική, είναι ένα νέο μέσο και πιστεύω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από μία σκέψη, από μία πτυχή. Είμαι πολύ υπέρ του, της προσεγγίσεως του δικού χάρτη που προτείνει ο εισηγητής και τη βούληση που δείχνει να ολοκληρωθεί το θέμα στην πρώτη ανάγνωση. Συμφωνώ με το χρονοδιάγραμμα. Νομίζω ότι όλοι έχουμε κάνει θυσίες, κάνουμε θυσίες για να μην βάλουμε μέσα όσα θα θέλαμε. Ίσως κρατήσαμε, συγκρατήσαμε κάπως τον εγωισμό και θέλουμε να είναι ολοκληρωμένη πολιτική και από την πλευρά των, ε, και στη Μεσόγειο. Να μην ξεχωρίζουμε κάθε χώρα. Πριν την ε, λήξη αυτού του ορίου θα πρέπει να ε, καθορίσουμε το επόμενο στάδιο με περισσότερους πόρους και με πειραματισμό που θα ξεκινήσει αυτή την περίοδο, Πρόεδρε. Μία από τι προτεραιότητε και κλείνω εδώ, που θα πρέπει να αναφέρουμε στη δραστηριότητα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον επόμενο χρόνο θα είναι η επαλήθευση, η, η εξακρίβωση του πώ εφαρμόζεται, πώ υλοποιούνται, πώ χρησιμοποιούνται οι πόροι που διαθέτουμε σε αυτή τη φάση, σε αυτό το στάδιο. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην κυρία Μπανίνη, θα ήθελα και εγώ να απευθύνω μια έκκληση δεν θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, γιατί μιλάμε για ολοκληρωμένη θαλάσσια περιοχή, για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε έχουμε και την Κελτική και την Ελλαδική θάλασσα, αλλά <laughs> δεν πρέπει να κολλάμε εκεί πέρα. Είναι ολοκληρωμένη η θαλάσσια πολιτική. Ας το έχουμε αυτό υπόψη. Είναι γενική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Μπενίνη, εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Επιτροπή σας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προσοχή που δίνετε και το έργο σας για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τον εισηγητή που είχε τόσο αγαστή συνεργασία με τους εκπροσώπους και των άλλων επιτροπών. Σίγουρα θέλουμε να αναπτύξουμε την πολιτική αυτή που είναι νεοπαγής, έχει μόνο τριετή ζωή και στηριχθήκαμε σε κάποιες προπαρασκευαστικές δράσεις και πιλωτικά προγράμματα και τώρα έχουμε μια νέα ευκαιρία για να αξιοποιήσουμε τις μέχρι τώρα προσπάθειές μας και να δούμε πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμη και πόσο φιλόδοξοι μπορούμε να είμαστε. Δεν θα πρέπει επίσης να μελούμε και να ξεχνούμε ότι στόχος τη ε, ολοκληρωμένη πολιτική δεν είναι να υποκαταστήσει τομεακέ ή κλαδικέ πολιτικές. Δεν πρόκειται να υποκαταστήσουμε ούτε την ενεργειακή πολιτική, ούτε θα αποπειραθούμε ε, να ε, έχουμε επικάλυψη κονδυλίων άλλων πολιτικών, της ενεργειακής, της αλλιευτικής, της περιβαλλοντικής πολιτικής. Βασικό μας έργο και καθήκον, γι' αυτό και το κονδύλιο αυτό είναι τόσο πενιχρό, τόσο περιορισμένο, είναι να δημιουργήσουμε κάποιες γέφυρες μεταξύ των διαφόρων πολιτικών, ώστε να υπάρχει μια συνειδητοποίηση του αντικτύπου των δύο αυτών πολιτικών στο περιβάλλον ε, της θάλασσας. Ο απότερος μας σκοπός είναι να προωθήσουμε μια αηφόρο χρήση των θαλασσών και των δραστηριοτήτων που ε, λαμβάνουν χώρα σε θαλάσσιο περιβάλλον. Θα ήθελα να δώσω κάποια απάντηση στην κυρία Φώστερ για την τροπολογία 7, για το κατά πόσο όρος implementation, εφαρμογή, ε, δημιουργήσει κάποια αμφισβήτηση της επικουρικότητας ή μιλούμε για εφαρμογή μόνο για τα κράτη-μέλη της περιοχής. Φυσικά, ναι και όχι ταυτόχρονα, γιατί ναι μεν αφορά τα κράτη-μέλη της περιοχής, αλλά μερικές φορές χρειαζόμαστε κάποιες κοινοτικέ δράσεις, δράσεις σε κοινοτικό επίπεδο, για να εξασφαλίσουμε αποτελεσματικότητά τους. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε κάποια δεδομένα, συγκέντρωση δεδομένων για την κατάσταση θάλασσας με συμβατό τρόπο και καλύτερη απορρόφησή τους και αξιοποίησή του από τα Εθνικά Στατιστικά Ινστιτούτα, θα πρέπει το έργο να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να είναι πραγματικά συμβατά αυτά τα δεδομένα. Το ίδιο ισχύει και για την ε, ανταλλαγή κάποιων δεδομένων για την ε, εποπτεία και παρακολούθηση. Χρειαζόμαστε κάποια συμφωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να εξασφαλίσουμε καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων αυτών από όλου του κλάδου και με παρόμοιο τρόπο σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Ναι, το βασικό άχθος της εφαρμογής ε, ε, καλύπτει τα κράτη-μέλη και φυσικά η αρχή της επικουρικότητας ε, περιτανεύει σε όλες μας τις δράσεις. Κύριε Κούν, θέσατε μία πολύ εύστοχη ερώτηση για το πώς θα εξασφαλίσουμε εφαρμογή των μακροστρατηγικών από τα κράτη-μέλη. Πώς θα το εξακριβώσουμε αυτό. Αυτό είναι ένα έναο έργο. Καταρχήν συγκεντρώνουμε κάποιες πληροφορίες από τα κράτη-μέλη και από τις ε, περιφέρειες ε, που δημιουργούν αυτή τη θαλάσσια λεκάνη και θεσπίζουμε δέσμοι των κατάλληλων δράσεων, συνεχίζουμε το διάλογο με τις ομάδες εμπειρογνωμών των κρατών μελών για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και στην ε, αρμόδια ομάδα εργασίας του Συμβουλίου και Έχουμε τακτικέ ενημερώσεις. Ένα από τα πλεονεκτήματα της ε, ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτικής και των ε, στρατηγικών που θα αναπτυχθούν στις θαλάσσιες λεκάνε, με βάση αυτή την ολοκληρωμένη στρατηγική είναι ότι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια συνέχεια στον, αυτόν τον εδαφικό σύνδεσμο με τα κράτη-μέλη. Και δεν μιλούμε μόνο για εδαφική και περιφερειακή πολιτική με βάση κάποιε ξεχασμένε συγκεκριμένε δράσει, αλλά θέλουμε να θεσπίσουμε πιο μακροπρόθεσμου στόχου οι οποίοι θα τη και κάποιε αναθεώρησει σε, διάφορα διαστήματα. Μην ξεχνάτε ότι ναι, μεν πρόκειται για μια νεοπαγή πολιτική, αλλά πιστεύουμε ότι θα αναπτυχθεί και θα αναδειχθεί πολύ περισσότερο στο μέλλον. Κύριε Κουμουτσάκο, έχετε να προσθέσετε κάτι. Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο με επικοδομητική διάθεση και με συγκεκριμένες ιδέες και απόψεις που θα με απασχολήσουν. Θα ήθελα να απαντήσω πρώτα απ' όλα σε δύο ανησυχίες που εκφράστηκαν. Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά το δούριο ύπο, πρέπει να σας πω ότι στην, στις επαφές μου με το Συμβούλιο αισθάνομαι ότι εγώ είμαι ο δούριος ύπος γιατί έχω και το know-how. Ως If you're seen as the Trojan horse, that's fine. Εντάξει, αν εσείς θεωρείτε τον εαυτό σας δούριο ύπο, κανένα πρόβλημα. Όσα ε, Έλλην μπορείτε να εκτιμήσετε το Συμβούλιο. not, not vice versa. Uh, regarding uh, Mrs. Εγώ θα είχα αυτό το ρόλο και όχι το αντίθετο. Σε ό,τι αφορά το παράπονο της κυρίας Μάισνερ για την συμμετοχή των συναδέλφων, απουσιάζει βέβαια η κυρία Μάισνερ, αλλά θα ήθελα να την καθησυχάσω, γιατί στην επόμενη φάση όταν θα ξανακαταρτήσω το κείμενο, θα περιλάβω και ένα πιλωτικό πρόγραμμα για μια θαλάσσια ευρωβινέτα που θα πρότεινα να συμπεριληφθεί στην ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Στο επόμενο συζήτηση λοιπόν θα έχουμε πολύ πιο αθρώα προσέλευση γιατί θα έχουμε ευρωβινέτα και στις θαλάσσιες μεταφορές. Και έρχομαι και στα πιο σοβαρά θέματα τώρα. Φαντάζομαι θα πρέπει να το ξεκαθαρίσετε με την κυρία Βάρτμαν Κόλ αυτό, κύριε Κουμουτσάκο. Το κείμενο, ο κανονισμό που συζητάμε σήμερα δεν είναι ένα πολιτικό κείμενο πλαίσιο. Έτσι, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ένα χρηματοδοτικό μηχαν... Ε, ένας χρηματοδοτικός κανονισμός είναι αρκετά τεχνικός και δεν θα πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε ως ένα πολιτικό κείμενο που όλα μπορούν να αναφερθούν. Ε, θα ήταν χαρά μου αν μπορέσω να το κάνω, αλλά θα ξεπεράσω και θα κινηθώ πέραν ε, της αποστολής που έχει το συγκεκριμένο κείμενο. Ε, να πω και εγώ για να είναι σε όλους σαφές ότι με την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική δεν χτίζουμε αχτές. Οι ακτές υπάρχουν, δεν επηρεάζουμε τις ακτές δηλαδή τις άλλες πολιτικές, προσπαθούμε να χτίσουμε γέφυρες. Επομένω, αυτό είναι ο στόχο και όχι να επηρεάσουμε άλλε επιμέρου πολιτικέ. Ε, όσον αφορά τι παρατηρήσει που ακούστηκαν πολύ γρήγορα για τον κύριο Μιλάνα, με απασχόλησε και εμένα πάρα πολύ και το ξέρετε ότι το συζητήσαμε αν μπορούμε να εξειδικεύσουμε περισσότερο τις δράσεις και ακόμα περισσότερο να ορίσουμε όριο δαπανών και όριο, όριο δαπάνες για κάθε δράση. Οι συζητήσεις που είχα, λεπτομερείς και ενδελεχείς, και φάνηκε και από την απάντηση της, του κυρίου Ρικέ όσον αφορά τον προπολογισμό, δείχνουν ότι θα ήταν μια πολύ δύσκολη, σχεδόν αδιέξοδη προσπάθεια. Αυτό ήταν ο λόγος που δεν αναφέρομαι ε, στο κείμενο παρουσία σα σε spending maxima κατά κατηγορία. Αυτή η διάσταση μεταξύ πολύ γενικού και πολύ ειδικού ε, ήταν αυτή που με απασχόλησε και στην πρόταση προσπάθησα να γεφυρώσω αυτές τις δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Ε, όσον αφορά στη Μεσόγειο, βεβαίως η Μεσόγειος είναι και δεν θα μπορούσατε να περιμένετε μια άλλη αντίδραση από έναν Έλληνα. Θεωρώ και εγώ ότι είναι η πιο σημαντική θάλασσα της Ευρώπης, όμως δεν μπορούμε να αγνοήσουμε άλλες θαλάσσιες περιοχές που για τα κράτη τα οποία βρίσκονται εκεί έχουν εξαιρετική σημασία. Αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει πόσο μικρό είναι το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Ε, όσον αφορά την ε, ανησυχία της κυρίας Μάισναρ για την τροπολογία 28, θα ήθελα απλώς να πω ότι είναι μια τυπική αναφορά που προκύπτει από την διαδικασία ε, των, ε, των delegated acts. Ε, για τον κύριο Τέιλορ, τα ETS όπως σας είπα, γενικά δεν είναι ένα πολιτικό κείμενο πλαίσιο, αλλά ένα τεχνικό θέμα, ένα τεχνικό κείμενο. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα μέσα. Ε, και, εν πάση περιπτώσει, έχω προσπαθήσει να λάβω πολύ σοβαρά υπόψη μου τις ευαισθησίες για το περιβάλλον και για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που είναι άλλωστε και δικές μου ευαισθησίες, αλλά δεν πρέπει, νομίζω, σε αυτό να προχωρήσουμε σε πολιτικές αναφορές για άλλους τομείς που θα υπάρξουν άλλα κείμενα τα οποία θα αναφερθούν ε, σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις όπως το ETS ή το CO2. Ε, τώρα, όσον αφορά την, ε, την παρατήρηση του κυρίου Βαντάλεν για την τροπολογία 17, ε, είναι ακριβώς αυτό ή προσπάθησα να αποτυπώσω αυτό που λέει και η Επιτροπή να μην υπάρχουν επικαλύψεις με άλλες πολιτικές. Ε, όσον αφορά τις γενικές εξαγγελίες, σας είπα ότι προσπάθησα να βρω ένα μέσον όρο. Οι πράσινοι λιμένες είναι κάτι το οποίο θα ακούω ότι θα κάνετε τροπολογία, θα πρέπει να το μελετήσουμε και να το δούμε. Δεν είμαι εξ αρχής απορριπτικός, αλλά είναι κάτι που πρέπει να δούμε. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ντομινίκ για την πολύ σαφή του τοποθέτηση όσον αφορά το δύσκολο και πολύπλοκο θέμα του προπολογισμού. Ε, στο Συμβούλιο ε, ακούω ότι υπάρχουν κράτη που σκέφτονται να πάνε στο, ε, στο reallocation of funds, αλλά είναι κάτι που θα περιμένω και να επιβεβαιωθεί και να το δω. Ε, κατά τα άλλα, ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις του και την κυρία Φώστερ και τον συνάδελφο τον κύριο Κούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 17 Μαρτίου. Ψηφοφορία στην Επιτροπή Μεταφορών θα λάβει χώρα τον Απρίλιο και ε, ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Ιουνίου. 17 λοιπόν Μαρτίου, προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κουμουτσάκο. Πάμε τώρα στην γνωμοδότηση για την έγκριση. Έγκριση τύπου και οπεδίες αγοράς δικύκλων και τρικύκλων οχημάτων, καθώς και τέτρα κύκλων. Ο κύριο Σίλερ είναι ο ημερογνώμονα τη Επιτροπή μα. Κύριε Ζήλα, παρακαλώ. Ναι, σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό, κύριε Ζήλα. Please. Thank you. Mr. Zila. Uh, ευχαριστώ. Λοιπόν, επειδή πάντα χρησιμοποιούμε την αγγλική γλώσσα στην προετοιμασία των εκθέσεων και συναντήσεις με τις ε, διαφορετικές ομάδες, δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο θα μπορούσα να σας εξηγήσω όλες τις λεπτομέρειες του φακέλου στην μετρική μου γλώσσα. Λοιπόν. Ε, ε, λοιπόν, η πρόταση της ε, Επιτροπής για τα οχήματα αυτά κατηγορίας ΛΑΜΝΑ συμπεριλαμβάνει ηλεκτρικά ποδήλατα, μοτοποδήλατα, γύκλες, τρίκρες, μοτοσυκλέτες, τετράκυκλες καθώς και μην οχήματα. Υπάρχουν ορισμένες απαιτήσει τεχνικές για να μειωθούν τα ε, επίπεδα των εμπομπών, να αυξηθεί η ασφάλεια, να υπάρχουν νέες ε, διοικητικές και τεχνικές απαιτήσει και να ε, απλουστευτεί το νομικό πλαίσιο. Ε, αν εξετάσουμε τα αριθμητικά στοιχεία όσον αφορά τον αριθμό των πόσων μοτοσυκλιστών και λοιπά σκοτώνονται στους δρόμους μας είναι 6.000 ο αριθμός αυτός σε όλους τους τύπους των οχημάτων και υπάρχει ένας υπολογισμός που λέει ότι 16% των ε, θανάτων στους δρόμους μας είναι οδηγοί των ε, οχημάτων αυτών, ενώ 2% ε, αποτελούν οι οδηγοί αυτοί στο σύνολο των οδηγών χρηστών των δρόμων. Το ποσοστό δηλαδή είναι τεράστιο. Και γι' αυτό μια από τις μιας προτάσεις είναι να είναι υποχρεωτική η πρόβλεψη των ε, συστημάτων ε, πέδησης αντιεμπλοκής ε, προηγμένων συστημάτων αντιλόκ και θα θέλαμε να διευρύνουμε την παλιά πρόταση γιατί καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο ήταν μέχρι στιγμή η διαπραγματεύση με την Κομισιόν και του ενδιαφερόμενους κύκλους. Εμείς στην Επιτροπή Μεταφορών θέλαμε να προτείνουμε κάτι αρκετά προκλητικό εδώ και αφορά την κατηγορία των ε, οχημάτων ε, της κατηγορίας L3εα1. Πρόκειται δηλαδή για μοτοποδήλατα με ταχύτητες πάνω από 80 χιλιόμετρα την ώρα. Και προτείνουμε να γίνει μια διάκριση το ανάλογο με το όριο ταχύτητας και να ζητήσουμε για την κατηγορία αυτή των οχημάτων που ξεπερνάνε τα 80 χιλιόμετρα υποχρεωτική επιβολή των συστημάτων πέδησης αντιεμπλοκής. Εάν δηλαδή τα οχήματα αυτά ξεπερνάνε την μέγιστη ταχύτητα των 80 χιλιόμετρων ανά ώρα. Πρέπει να είναι υποχρεωτική η... υποχρεωτικό εξοπλισμό. Γιατί μερικά από τα ταχύματα αυτά φτάνουν μέχρι τα 110 ε, χιλιόμετρα την ώρα. Γιατί στο κάτω-κάτω αυτό που σκοτώνει στους δρόμους δεν είναι η ισχύ του κινητήρα, αλλά η ταχύτητα με την οποία κινείται το όχημα. Γι' αυτό θέλουμε την τροποποίηση αυτή. Επίση στα συστήματα πέδηση αντιεμπλοκή συζητιέται συχνά το θέμα του κόστους. Συνήθω δεν είναι πάρα πολύ ακριβό το σύστημα. Έχουμε στοιχεία από τους πολιτές 100 με 200 ευρώ στοιχεία από τους κατασκευαστές ε, της τάξης των 200-400 ευρώ ανά όχημα. Αλλά αυτό τι σημαίνει. Ένα τέτοιο μοτοποδήλατο, μια τέτοια μοτοσυκλέτα ε, έχει μια διάρκεια ζωής 10 ετών, το κόστος είναι 40 ευρώ το χρόνο. Το ίδιο έχει αυξηθεί και η τιμή των καυσίμων σε ένα χρόνο. επιχείρημα του κόστους λοιπόν κατά δεν είναι επαρκές. Η άλλη ε, σημαντική τροποποίηση είναι να συμπεριληφθούν τα οχήματα για χρήση εκτός του δρόμου. Υπάρχουν διαφόρων τύπων. 800.000 υπολογίζεται ότι υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συχνά χρησιμοποιούνται και στους δρόμους, όχι μόνο εκτός δρόμου και γι' αυτό θα πρέπει να ε, πληρούν ένα ελάχιστο επίπεδο προτύπων ασφαλείας. Στο τρίτο θέμα είναι οι προδιαγραφές επιδόσεων στους δοκιμές πρόσκρουσης. Ε, πολλά από τα οχήματα που συμπεριλαμβάνονται να στην οδηγία δεν έχουν καθόλου δοκιμές πρόσκρουσης. Είναι λοιπόν για το μέλλον αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ ευάλωτα και οι οδηγοί τους βέβαια και εκείνοι που ταξιδεύουν σε αυτά είναι ευάλωτοι. Επίσης θέλω να συχθεί μια νέα υποκατηγορία για τα, τις μοτοσυκλέτες Enduro και Trial. Γιατί συνήθως χρησιμοποιούνται για εκτός δρόμου, αλλά καμιά φορά χρησιμοποιούνται και στους δρόμους. Και στην περίπτωση αυτή πρέπει βέβαια, όπως είπαμε, να τηρούν ορισμένα τεχνικά πρότυπα ασφαλείας. Και όσον αφορά τις ε, εκπομπές και το χρονοδιάγραμμα, στις γενικές γραμμές συμφωνούμε με την πρόταση της Κομισιόν. Το μόνο θέμα που παραμένει ανοιχτά είναι το επίπεδο ευρώ 4 για τα μοτοποδήλατα τα οποία πραγματικά μολύνουν πάρα πολύ αν δει κανένα πόσα χιλιόμετρα ε, χρησιμοποιούνται και πόσες εκπομπές έχουν. Και γι' αυτό θέλουμε να εισαχθεί αυτό το πρότυπο Ευρω 4 για τα μοτοποδήλατα τρία χρόνια νωρίτερα, δηλαδή το 2014 ήδη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ζήλα, ο κύριος Σίγκεντς. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε Συμφωνώ σχεδόν με τα πάντα που είπε ο κ. Ζήνα, έκανε έξοχη δουλειά. Συνάθρισε 14 εκθέσεις, 14 οδηγίες. Αυτό χρειαζόμαστε. Μεγαλύτερη ενοποίηση κειμένων, περισσότερη ενοποίηση, κυρίως στον κατασκευαστικό τομέα. Εκεί πρέπει να κινηθούμε, προς τα εκεί. Αν υπάρχουν διαφορετικές οδηγίες όσον αφορά την κατασκευή αγαθών και οχημάτων, το ένα ασχολείται με τους ήχους, το άλλο με εκπομπές, το άλλο με ασφάλεια και το καθεξής, Νομίζω ότι έκανε έξοχη δουλειά, όπως ε, είπε, σκοπός είναι να συναθρήσουμε όλα αυτά τα στοιχεία μαζί και να μειώσουμε τις εκπομπές, να βελτιώσουμε και την οδική ασφάλεια. Και τέλος, κάτι εξίσου σημαντικό, να λάβουμε υπόψη τις νέες τεχνολογίες και εποπτεία, που είναι, είναι μια λέξη που αναφέραμε στην άλλη έκθεση. Εποπτεία, ο έλεγχος είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ζωτική σημασία ούτως ώστε να μην εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση οχήματα από χώρε, π.χ. από την Κίνα, που υπολείπονται των προδιαγραφών, δεν συμμορφώνονται με τα διάφορα πρότυπα που έχουμε θεσπίσει για του δικού μα κατασκευαστέ οχημάτων. Πολύ καλή η προσέγγιση. Και είναι καλό που αντιστάθηκε στι πιέσει που το ασκήθηκαν από τι κατασκευαστικέ εταιρείε, διότι έχουν διάφορα συμφέροντα. Θέλουν να υπάρχει χαλαρότης. Και έθεσε όρια ασφαλείας προδιαγραφές και το ABS, το αυτόματο σύστημα τροχοπέδησης είναι κάτι που συμπεριλαμβάνεται. Καμία τροπολογία του ΕΛΚ θα εκτοχιάσει το έργο του συγητού. Και όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, Έχουμε νομίζω δική μου συμφορία στο, τον Ιούνιο στην Επιτροπή και το Σεπτέμβριο στην Ολομέλεια. Θα συνεργαστούμε για να πετύχουμε το βέλτιστο δυνατό ε, αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτά έχω να πω και συγχαρητήρια στον εισηγητή. Πρόεδρος, ο κ. Αλκαντράουι έχει τον έχω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μόλις έμαθα ότι η σκιώδη συγγήτριά μας, η ε, σήμερα. Θα την αντικαταστήσω εγώ και θα εκφράσω με δύο λόγια τη θέση της ομάδας μου. Χαίρομαι για την προσπάθεια πλούστευσης της νομοθεσίας, συγχώνευσης των νομοθετικών δράσεων σε ένα κανονισμό που θα πλουστεύσει τις διαδικασίες για τη θέση εμπορία και επιστοποίηση αυτών των οχημάτων. Πιστεύω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε ζητήματα ασφάλειας και να ενισχύσουμε την ασφάλεια των μοτοσυκλετιστών, που είναι ομάδα προτεραιότητας για τους ευάλωτους χρήστες ε, την επόμενη δεκαετία. Γενικώ είμαστε υπέρ της ε, συμπερίληψης του συστήματος ABS ε, αντιεμπλοκής, δηλαδή τροχών κατά την πέδηση σε όλες τις κατηγορίες, αλλά θέλουμε περισσότερη ενημέρωση κατά το πόσο το ABS είναι χρήσιμο σε κάποιες μοτοσυκλέτες low performance και αν κάτι τέτοιο θα συμβάλλει στον περιορισμό των ατυχημάτων. σε ό,τι φορά την αυτόματη, το αυτόνομα όνομα των ε, του, των, φωτών για όλα τα οχήματα νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να δούμε το θέμα της ε, προσαρμογής. Επίσης ε, θα πρέπει να εξετάσουμε περαιτέρω την πρόταση για τη δημιουργία νέων κατηγοριών για, τις, για, για τα οχήματα παντός εδάφους και να προσθέσουμε νέα στοιχεία ασφάλειας και προδιαγραφές για προστασία, ε, ταχύτητα, εφίους προσαρμογής ταχύτητας και επίσης το θέμα της κατάρτισης και της υποδομής ε, για τις μοτοσυκλέτες. Ε, όταν μιλούμε για την ασφάλεια για τις μοτοσυκλέτες είναι πολύ σημαντικό, δεν θα πρέπει να το ξεχνούμε και αυτό. Πάντως πιστεύω ότι μπορούμε να διαμορφώσουμε μια καλή γνωμοδότηση της Επιτροπής μας και υποστηρίζουμε πλήρως το έργο του εισηγητού. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στέρξ. Ευχαριστώ. Και εμείς πιστεύουμε ότι η έκθεση είναι πολύ καλή και όπως είπε και ο συνάδελφος συμφωνούμε με τις αδρές γραμμές του εγγράφου. Έρχομαι σε κάποιες συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Η τροπολογία 2 για την οδική ασφάλεια είναι γέννη. Πολύ καλή. Θα πρέπει επίση να επιστήσουμε την προσοχή ε, στο θέμα της κατάρτισης που είναι πολύ πιο σημαντική για τα δίτροχα και τα τρίτοχα τράτροχα παρά για τα οχήματα σχεδόν. Και θα πρέπει να δούμε και το θέμα της ασφάλειας των μοτοσυκλετιστών αν έχουμε τροπολογία για την, ασφάλεια, για την οδική ασφάλεια, θα πρέπει να περιλαμβάνει μια τέτοια τροπολογία και την κατάρτιση και τις υποδομές. Γιατί στις υποδομές, οι υποδομές είναι θεμελιώδες ε, υπόθεμα για τη χρήση των ε, μοτοσυκλετών. Θα μπορούσαμε να ζητήσουμε και αμεσότερη ε, εφαρμογή ορισμένων μέτρων ασφάλειας. Ας το σκεφτούμε και αυτό. Συμφωνώ και με τον Σαΐντ για το θέμα το κατά πόσο είναι δυνατόν να προβλέψουμε αυτόματο άνοιγμα των φώτων και για τις μοτοσυκλέτες. Ίσως θα μπορούσαμε να σκεφτούμε αυτόματους ε, διακόπτες που ανάβουν. Ευχαριστώ κύριε Λίχτεμπερμα. Εκτός μικροφώνου. Okay. Uh, ich möchte mich einem Punkt Λοιπόν, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα σημείο και συγκεκριμένη διάκριση ανάμεσα σε ένα πραγματικό ποδήλατο, ένα, μια πραγματική μοτοσυκλέτα και όλα αυτά που υπάρχουν διάμεσα. Γιατί υπάρχουν και ποδήλατα ηλεκτρικό ε, κινητήρα που κινούνται με ταχύτητα κάτω των 25 χιλιόμετρων ώρα. Εάν το αποζητάμε από αυτούς τα ίδια μέτρα ασφαλείας όπως από άλλους, τότε είμαστε πολύ άνηση γιατί θα πρέπει να αναμετρηθούν με κατηγορίες με τις οποίες δεν έχουν καμία σχέση όσον αφορά τις εκπομπές ή το θέμα της ε, ταχύτητας κλπ. Θα ήταν ίσως καλό να σκεφτούμε μήπως αυτά θα πρέπει να εξαιρεθούν αυτά τα ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα που δεν είναι μόνιμη χρήση κινητήρα για τα εν λόγω οχήματα. Ε, και υπάρχει σημαντική διαφορά όσον αφορά και την χρήση και τον τρόπο χρήσης και τις αποστάσεις. Όταν εγώ ήμουνα φοιτήτρια πήγα με ένα μοτορίνο στην Ιταλία και πέρασα 600-700 χιλιόμετρα. Δεν θα μπορούσα να το κάνουμε αυτό όμω με ένα ε, ποδήλατο με βοηθητικό κινητήρα, γιατί αυτά προβλέπονται μόνο για μετακινήσεις μέσα στην πόλη κλπ. Γι' αυτό πιστεύω ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές και θα ήταν καλό να μην τα συμπεριλάβουμε γιατί θα υπήρχε πολύ με έντονο διοικητικό άχθος για κάποιες κατηγορίες οχημάτων χωρίς να έχουμε ανάλογο αποτέλεσμα όσον αφορά την ασφάλεια ή την μείωση των εκπομπών. Και κάτι άλλο με την ενεργοποίηση των φανών κατά τη διάρκεια της ημέρας. Φοβούμε ότι υπάρχει διαφοροποίηση ανάλογα με το πόσο φως υπάρχει κατά τα άλλα γύρω. Εμείς έχουμε μελέτες στην Αυστρία σε δεν οδηγεί σε βελτίωση της ασφάλειας το γεγονός ότι η φανή είναι αναμένη την ημέρα. Εμείς δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κάτι που κοστίζει πολύ ενέργεια χωρίς να αποδίδει το ευκταίο αποτέλεσμα. Μου φαίνεται ότι όλη αυτή η ιδέα με τον ε, φως κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι ένα σπιράλ που προχωράει. Άρχισε με τα αυτοκίνητα, τότε θα πρέπει να ισχύει αυτό και για τα δίτροχα και κάποια στιγμή θα είναι υποχρεωτικό και οι πεζοί και τα παιδιά να είναι φωτισμένοι για να μπορούν να τους βλέπουν στο δρόμο. Παράλογο κατά τη γνώμη μου. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Mm. Θα ήθελα και εγώ να πω δύο λόγια. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την έκθεσή του που ήταν πάρα πολύ ε, ενδιαφέρουσα για τα δίτροχα, τίτροχα και τετράκλατα αυτά ε, ε, οχήματα. Νομίζω πραγματικά ότι τα ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα θα πρέπει να εξερθούν. Εγώ τα βλέπω συνήθως στην Ολλανδία. Mm. Είναι ας πούμε ένα ποδήλατο για τους τεμπέληδες κατά κάποιο τρόπο αυτό. Ναι, πραγματικά δέχομαι ότι είναι τόσο χαμηλή απόδοση που δεν αξίζει το λόγο να συζητώ. Εκεί που υποστηρίζομαι στον εισηγητή είναι όταν περάσουμε στα μοτοποδήλατο που τα βλέπουμε πολύ στη Ρώμη Φερρυπής και στη Μεσόγειο πάει κανένας ε, <laughs> στο μοτοποδήλατο με σότς και σαγιονάρες ξέρετε τι εννοώ ε, αυτά τα οχήματα θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ένα σύστημα ε, με πέδηση αντιεπλοχής γιατί το 20% των δυστυχημάτων με τα οχήματα αυτά θα μπορούσαν να έχουν επιφευθεί εάν είχαν συστήματα πέδησης αντιεπλοχής. Είναι θέμα λοιπόν οδικής ασφάλειας αυτό και δικαίως ο εισηγητής αναφέρθηκε στο ότι οι παραγωγοί, οι κατασκευαστές αναφέρονται στο θέμα του κόστους. Εγώ αναρωτιέμαι πάντα, μια ζωή πόσο κοστίζει. Αυτό είναι. Λοιπόν, όλα αυτά τα σκούτερ, τα παπάκια, τα ξέρετε τι λέω. Όλα αυτά τα ποδήλατα θα πρέπει να έχουν ένα σύστημα του πέδησης αντιπλοκής. Και κάτι άλλο. Η κυρία αναφέρθηκε σε αυτό. υπήρχε η αντίθεση να υπάρχουν οι φανή ημέρας αναμένη στα αυτοκίνητα για να είναι αναμένοι στα δίτροχα και να μπορούν να ξεχωρίζονται τα δίτροχα στο δρόμο. Έχουμε διάφορα παραδείγματα τρελών οδηγών όλοι. Εμείς έχουμε ένα δρόμο στη δική μου εκλογική περιφέρεια που είναι το χειρότερο σε αφορά τα δυστυχήματα. Γιατί έχει πάρα πολλές στροφές ε, και το χρησιμοποιούνται οι μοτοσυκλετιστές για αγώνες. Και καταφέρνουν να θερμάσουν να σκοτωθούν εκεί. Λοιπόν, πολλά από τα δυστυχήματα που σχετίζονται με μοτοσυκλέτες δεν οφείλονται στη μοτοσυκλέτα αλλά στο μοτοσυκλετιστή. Και αυτό θα είναι κάτι που θα πρέπει να το έχουμε κατά Μετά, ξέρω ότι όλοι ανησυχείτε μήπως κάποια στιγμή και οι πεζοί θα πρέπει να έχουν φώτα ή κάτι. Να σας πω, ε, σε ορισμένες ε, ε, υπαίθριες περιοχές που δεν υπάρχουν φώτα στον δρόμο, δεν είναι κακή ιδέα να έχει ένα φακό στο χέρι του, στο κεφάλι του ο πεζός. Εγώ θα ε, έλεγα ότι θα ήταν καλό ποδηλάτες να έχουν φώτα. Γιατί υπάρχουν πολλοί ποδηλάτες που δεν έχουν φώτα στα ποδήλατά τους. Απίθανο. Και μετά απορούν γιατί τους χτυπάει το αυτοκίνητο μέσα στη μέση της νύχτας. Αυτοί σωστά πρέπει να φοράνε ένα φακό στο κεφάλι. Από την άλλη μεριά βέβαια όσο καλή νομοθεσία και αν έχει κανένας, εάν κάποιο ηλίθιος ε, ε, ανεβαίνει στη μοτοσυκλέτα θα σκοτωθεί. Τι θα κάνουμε. Η έκθεση πάντως είναι πολύ καλή και οπωσδήποτε υποστηρίζω την ε, γραμμή που παρουσιάσατε. Ιδιαίτερα τα συστήματα πέδησης αντιεμπλοκής. Μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό αυτό. For the commission, Mr. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Greenley. Αν έκανα λάθος το όνομά σας, ζητώ συγγνώμη, αλλά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Λέμε έτσι, πρωί είναι ακόμα. Α, δίκιο έχετε, δίκιο έχετε. Ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα να προβούμε σε κάποια σχόλια και να δώσουμε κάποιες πληροφορίες. Γιατί προτείναμε αυτό που έχετε μπροστά σας. Να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή καταρχάς διότι είδαμε ότι υπάρχουν πολλές λογικές τροπολογίες που μπορούμε να υποστηρίξουμε όμως υπάρχει κάτι που ανέφερε. όπου η πρόταση είναι εκεί για να τροποποιήσει το πώς τοποθετούνται στην κατηγορία L3-1α της κατηγορίας των μοτοποδηλάτων με χαμηλή ισχύ σύστημα πέδησης αντιμπλοκής είναι για να κάνουμε διαφοροποίηση μεταξύ των οχημάτων. Στην αξιολόγηση συνεπιών που κάναμε, δικαιολογούνται διάφορα πράγματα που προτείναμε. Ερευνήσαμε διάφορε παραμέτρου για να ξεχωρίσουμε τα οχήματα. Η ταχύτητα των οχημάτων είναι κάτι εύκολα μετρήσιμο, ξυπακούτε. Δυσκολότατη διαφοροποίηση όμως εντός υποκατηγοριών των, των μοτοποδηλάτων που πηγαίνουν με, με χαμηλή με μικρό κινητήρα τα οχήματα που πάνε με ταχύτητα μεγαλύτερα από 80 χιλιόμετρα την ώρα από εκείνα που έχουν ταχύτητα μικρότερα από 80 χιλιόμετρα την ώρα. Άρα βρήκαμε κοινά κριτήρια ανάμεσα στην οδηγία για την άδεια οδήγηση και τις προσέγγιση που ακολουθούμε για τις υποκατηγορίες. Έχουμε κατηγορίες 1α, 1, α 1 β και 1γ και αυτά συνδέονται και με την οδηγία για την άδεια οδήγησης. Αν κάποιος έχει άδειο οδήγηση για μοτοσυκλετα α Α1, τότε πρέπει να συμμορφώνεται με προδιαγραφές ο κατασκευαστής και θα πρέπει να θυγραμίζεται. Θα πρέπει ο τελικός χρήστης να ξέρει ότι αυτά τα οχήματα θα έχουν σύστημα πέδησης, σύστημα αντιεμπλοκής, είναι κατηγορίας Α1 και όλα τα ε, οχήματα που είναι πάνω από 125 κυβικά και πάνω από 11 κιλοβάτ θα έχουν σύστημα αυτό αντιμπλοκής. Προσπαθήσαμε να πετύχουμε διάφορους στόχους. Θέλαμε να πετύχουμε απλούστευση και βελτίωση για το περιβάλλον και για την ασφάλεια. Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο. Και να συμπεριλάβουμε και διάφορους μηχανισμούς εποπτείας και ελέγχου της αγοράς. Προσπαθούμε να εξορροπήσουμε τα διάφορα μέτρα που προτείνονται Κάθε μέτρο έχει κάποιο κόστος και για τους κατασκευαστές. Στην πρότασή μας προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε λογική προσέγγιση. Και δεν ξέρουμε αν θέλετε και περαιτέρω υποδιαίρεση. Για τα ηλεκτρικά ποδήλατα, σχόλιο. Τι προτείνουμε. Προτείνουμε αυτό που ισχύει. Υπάρχουν κάποια ποδήλατα που εξαιρούνται από την ομοθεσία. Δεν αλλάζει αυτό. Υπάρχουν κάποια ισχυρά δίκυκλα που συμπεριλαμβάνονται και με την πρότασή μας προσπαθούμε να διευκρινίσουμε αυτό. Δηλαδή τα ισχυρά δίκυκλα, τα ισχυρά ποδήλατα και προτείνει η βιομηχανία φτάσει και σε ισχύ επί 16 και εκεί να δούμε ποιες είναι οι απαιτήσει. Αυτά ήθελα να υπογραμμίσω και να θέσω στην προσοχή σας. Πριν μιλήσεις, Ρόμπερτ, ζητώ συγγνώμη που με τις θέσεις του Προέδρου. 125 κυβικά είναι πολύ μεγάλη ισχύ για συστήματα αντιεμπλοκής. Ό,τι είναι πάνω από 49 κυβικά θα πρέπει να έχει σύστημα αντιεμπλοκής στην πέδηση δίνεται φωνικά εργαλεία στον κόσμο και δεν τους προστατεύετε. Τα 125 κυβικά αποκλείονται. Όποια και, ό,τι και να λέει αξιολόγηση συνεπιών, σκασίλα μου. Εγώ θεωρώ ότι είναι ανόητο αυτό. Συγγνώμη, Ρόμπερτ, αν έχεις κάτι να πεις. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους έλαβαν το λόγο και από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουμε διαπραγματεύσουμε του οικειώδει συλλογητέ προκειμένου να καταλήξουμε συνενετικέ λύσει. Πάντω, σα ευχαριστώ για την υποστήριξη. Χαίρομαι για την εμπειρογνωμοσύνη τη Ευρω... Ευρωπαϊκής Επιτροπής να βρούμε τα σωστά κριτήρια για κάθε κατηγορία. Και εγώ έχω ανάμεικτα συναισθήματα, γιατί η αρχική μου πρόταση ήταν όριο ταχύτητα, υποκατηγοριοποίηση με βάση το όριο ταχύτητα. αλλά ίσω αυτή δεν είναι η καλύτερη λύση. Αλλά έχω εμπιστοσύνη ότι θα βρούμε καλή λύση σε ό,τι αφορά την, το αυτόματο άναμα των φανών. Δεν, δεν μπορούμε να σταματήσουμε τα αυτοκίνητα να κάνουν κάτι που κάνουν ήδη. Και θα ήταν ε, περίεργο να πετούμε από τα μοτοσυκλέτες κάτι που δεν απαιτούμε από τα αυτοκίνητα. Στις σκανδιναβικές χώρες είναι υποχρεωτικό για όλη τη χρονιά, ακόμη και το καλοκαίρι, όχι μόνο για το χειμώνα που έχει λίγο φως. Και λειτουργεί θαυμάσια το σύστημα και βελτιώνει την κατάσταση. Είναι υποχρεωτικό το άναμα των φανών, συνέχεια. Τώρα, στην υπόλοιπη Ευρώπη, μεταξύ τη ημέρα και τη συνήθεια, υπάρχει ένα διάμεσο ε, επίπεδο φωτισμού. Θα πρέπει να έχουμε ε, και για τους ε, Ποδηλάτε ακόμη και για τους πεζούς ε, κάτι τέτοιο υποχρεωτικό. Γιατί όταν περπατάει κανείς, όχι στον δρόμο, και στην άκρη του δρόμου να περπατάει, διατρέχει τον κίνδυνο να το χτυπήσει αυτοκίνητο. Μιλάμε για μια νέα γενιά ευκαιριών για το πώς μπορεί κανείς να ανάβει τα φώτα και τη μέρα. Το πρόβλημα του ποδηλάτε είναι ότι υπάρχει υποχρεωτική νομοθεσία. Οι ποδηλάτε στην καταστρατηγού δεν εφαρμόζουν οι φυστάμενε διατάξει. Ο κύριο Χιγίνη. Ξέρω για την εμπειρία της Αυστρία αλλά στον Καναδά η ε, υποχρεωτική, το υποχρεωτικό άνομα των φανών και τη μέρα μείωσε κατά 10 τα ατυχήματα, τα τροχαία ατυχήματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει στάνταρ αυτό και έχει και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, είτε πρόκειται για αυτοκίνητο, είτε πρόκειται για δίτροχο, για τρίτροχο. Θα ήθελα να σχολιάσω αυτή την παρατήρηση. Εξαρτάται από το πού το εφαρμόζουμε. Στις μεσογειακές χώρες, για παράδειγμα, ή στις νότιες χώρες, έχουμε πολύ περισσότερο φως, οπότε δεν βοηθά και πολύ το άναμα των φανών. γιατί δεν υπάρχει και το θέμα της ε, ομίχλης που επηρεάζει. Και σας παρακαλώ να μην καταλήξουμε να υποχρεώνουμε τον πεζό να φοράει κράνος ή να φοράει και ειδικό μπουφάν ε, για να προστατεύεται όταν περπατάει. Αυτό είναι ακριβώς που δεν θέλουμε. Γιατί Αν θέλουμε να προστατεύσουμε τον πιο αδύναμο ε, κρίκο στις μεταφορές, φυσικά πάντα είναι εκτεθειμένος, γιατί αν τον χτυπήσει αυτοκίνητο, ό,τι και να φοράει, πάλι θα βρεθεί χαμένος ο πεζός. Ναι, μερικές φορές, αν κανείς περπατάει σε αγροτικούς δρόμους που δεν είναι φωτισμένοι, καλό είναι να φοράει ένα φακό στο κεφάλι όπως έχουν ε, πολλές φορές στο, στο ναυτικό, αλλά αυτό είναι για την προσωπική ασφάλεια του καθενό. Πάντως, είναι γεγονός ότι οι ποδηλάτες έχουν απέτηση και σωστά βέβαια να τη χάνουν προστασία, να του σέβονται οι υπόλοιποι χρήστε του δρόμου, αλλά δεν έχουν μόνο δικαιώματα οι ποδηλάτε, έχουν και υποχρεώσει και υποχρεούνται όταν οδηγούν τη νύχτα να φέρουν κάποιο φω για να του αναγνωρίζουν οι υπόλοιποι οδηγεί. Ευχαριστώ. 25 Μαρτίου λήγει η προθεσμία για τις τροπολογίες. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας το Μάιο. Σας ευχαριστώ. Διακοπή προς το πάρο γιατί ολοκληρώσαμε την πρωινή μας συνεδρίαση. Θα επανέλθουμε στις 3 για την ανταλλαγή απόψεων με τον καλό μας φίλο κύριο Γαζεμβόφσκι το συντονιστή για τα λειτουργικά τμήματα ενέργειου χώρου. Ραντεβού στις 3.